Έχουμε απαρτία, μπορούμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Μια ανακοίνωση των αποφάσεων που πήραμε χθες το βράδυ στους συντονιστές. Σχετικά με τη δικασία των ακροάσεων των επιτρόπων, των επιτρόπων για τις επόμενες εκλογές. Τι κανόνες θα ισχύσουν. Θα απαντήσω σε αίτημα του Προέδρου του Κοινοβουλίου του κανονισμού σχετικά με το πώς θα δικαθίσταται ένας αντιπρόεδρος στην περίπτωση που υπάρξει μία παρέτηση για κάποιο λόγο αν χειρεύσει η θέση του αντιπρόεδρου προτάθη να δοθεί εντολή στο τμήμα ερευνών να κάνει μια μελέτη σχετικά προεφθά θύνουσα αναλογικότητα, το μαθηματικό τύπο που θα μας επιτρέψει μάλλον επ' αυτού θα έχουμε μια πρόταση επ' αυτού είχαμε και μια πρόταση DAF ε, μια πρόσκληση προς μαθηματικούς από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Μια αντιπροσωπεία της αντιπροσωπείας θα πάει στην Ουγγαρία 9 και 10 Δεκεμβρίου. Οι συντονιστές προτείνουν τρεις βουλευτές από το ΕΛΚ, δύο από το Συσιαλιστικό Κόμμα και ένα από κάθε μία από τις άλλες ομάδες. Ένα άτομο. Φυσικά οι Ούγγροι βουλευτές δεν θα τους ε, αφήσουμε απ' έξω αυτοί άσχετα με τον αριθμό που ορίσαμε μπορούν να πάρουν μέρος. Το 2011 προετάθησαν επισκέψεις με αντιπροσωπεία στην Ιταλία, Ρώμη και Φλωρεντία, στην Αγγλία, Λονδίνο και Κέμπριτζ, στην Πολωνία, Βαρσοβία και στο δεύτερο εξάμεινο στη Θανία. Το 2011 οι συντονιστές προτείνουν στις 26 Ιανουαρίου ακρόαση για τα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έγιναν και άλλες προτάσεις αλλά δεν ε, εγκρίθηκαν προς το παρόν. Θα δούμε αν θα οριστεί αυτή η ακρόαση για τις 26 Ιανουαρίου. Με τον πρόεδρο Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής, ζητάμε να συμμετάσχει στην συνεδρίαση στις 29-30 ε, Νοεμβρίου με ανταλλαγή απόψεων για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, ιδιαίτερα στον αφορά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Και θα... Επειδή ο, ο, ε, ετέθη ερώτηση προς τον πρόεδρο Μπαρόσο να αλλάξει τη μέθοδο που εφαρμόζεται Ζητάει δηλαδή το Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο Μπαρόσο να εφαρμόσει το άρθρο 87 του κανονισμού και μην αναφέρεται σε νομοθεσία για την οποία δεν έχουν τεθεί ερωτήματα. 18 Οκτωβρίου η επόμενη συνάντηση των συντονιστών για να συζητήσουμε τι συνέχεια θα δοθεί στην έκθεση DAF στο ενιαίο εκλογικό σύστημα. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε για την πρωτοβουλία πολιτών και καλούνται να παρουσιάσουν το σχετικό σχέδιο έκθεσης όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα μπορούσαμε να δούμε εδώ το σημείο 6 της ημίρης διάταξης που προέβλεπε την έγκριση του χρονοδιαγράμματος για την Επιτροπή για το 2011. Δεν υπήρξε αντίρρηση της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν και εδώ αντιρρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα όπως προτείνεται. Στις ανακοινώσεις αυτές σχόλια. Όχι. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η πρωτοβουλία των πολιτών. Πρωτοβουλία Πολιτών. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε τη συνάντηση με εκπροσώπους των εθνικών κομμάτων, των εθνικών ε, κοινοβουλίων. Σήμερα, με βάση την ε, πρόταση της εισηγήτριας Γκουρμάη και Λαμασούρ, καλέσαμε δύο προσωπικότητες που στο παρελθόν ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Είναι ο καθηγητής Γιούργεν Μέγερ, που έχει υπάρξει Γερμανός βουλευτής και ήταν ο κύριος υποστηριχτής και αυτός που προώθησε στα πλαίσια της συντακτικής της πρωτοβουλίας πολιτών και την δόκτωρα Σίλβα Ιβον Κάουφμαν, ευρωβουλευτής σε δύο θητείες της Επιτροπής μας και ήταν συγγήτρια στην Επιτροπή την Συνταγματική για τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε μέσω των δύο αυτών προσωπικότητων. Πριν σας δώσω όμως το λόγο στους δύο προσκεκλημένους, παρακαλώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκουρμάη, να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που με τον συνεισηγητή μας, Λαμασούρ, μπορούμε να συναντηθούμε με τους δύο εμπειρογνώμονες, την Σίλβια Κάφμαν, που είναι και η μητέρα ουσιαστικά αυτής της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Χαίρομαι που βρίσκεται εδώ. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και από αυτή τη θέση Πιστεύω ότι έδωσε μεγάλη όθηση στην πρωτοβουλία αυτή. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα και θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της. Προετοιμάζοντας την έκθεση αυτή, είχα την τύχη να συναντήσω αρκετούς εμπειρογνώμονες και με την Σίλβια συναντήθηκα. και με τον ε, Αλέ που είναι δικός μας συνάδελφος ε, συναντήθηκα αρκετές φορές που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ξεκινήσαμε έτσι την διαδικασία εκπόνησης της έκθεσης αυτής. Συναντηθήκαμε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, πάνω από 100 συναντήσεις κάναμε μαζί τους και προσπαθήσαμε να τους ε, πούμε και τις δικές μας ιδέες, να τους εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα εδώ και να συλλέξουμε εμπειρία από ολόκληρη την Ευρώπη. Φυσικά η Επιτροπή μας έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ε, νομίζω ότι τελικά η έκθεση αυτή ε, έχει μια ισορροπία και ο κύριος Έφνερ βοήθησε πολύ στην ομάδα τελικά είμαστε δύο γυναίκες και δύο άντρες. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο αχέγγυο για να οδηγηθούμε σε μια καλή έκθεση. Μπορούμε να έχουμε μετά συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Νοέμβριο μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, αλλά είναι δεύτερη φορά που εδώ σε αυτή την Επιτροπή το συζητάμε. Έχουμε και ακροάσεις κάθε τόσο και Πιστεύω ότι στα τέλη του Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και θα μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη ανάγνωση, αν όλα είναι εντάξει, τη βδομάδα που αρχίζει 13 Δεκεμβρίου. Έτσι θα δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχει μεγάλη βούληση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προσφέρουμε στους πολίτες μία πρωτοβουλία πολιτών φιλική προς τους πολίτες. Βέβαια, χρειάζονται οργανωτικά ζητήματα. Πολλές φορές έχουμε ιδέες που μας έρχονται από τις περιφέρειες, είναι τοπικού χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι μόνο 42% των πολιτών πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες ε, ευρωεκλογέ. Ας φροντίσουμε λοιπόν να δώσουμε σε όλους τους πολίτες οι ίδιες ευκαιρίες ώστε να μπορέσουν όλοι να έχουν πρόσβαση στο software και στην ε, πληροφόρηση. Αν έχουμε λιγότερο από ένα εκατομμύριο ε, υπογραφές, έχουμε 900.000, τι θα κάνουμε. Είναι ένα ερώτημα. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι, εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες, να τους εξηγήσουμε ότι θέλουμε τη συμμετοχική δημοκρατία και ότι θα δώσουμε σημασία στα αιτήματά τους. Ο στόχος μας είναι κοινό. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες πρωτοβουλίες πολιτών και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να καταλάβουν τις ρυθμίσεις, να καταλάβουν τι κάνουμε εμείς εδώ και να μικρύνουμε την απόσταση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο πολίτη. Εμείς ξέρουμε πόσο χρήσιμη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη να το εξηγήσουμε και στους πολίτες. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να οδηγηθούμε σε νομοθεσία. Επαναλαμβάνω ότι θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να ενημερωθούν καλύτερα για το νέο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για νομοθεσία. Θέλουμε να είναι ένα ισχυρό μέσο δημοκρατικό, να μην γίνονται καταχρήσεις, να χρησιμοποιείται για ευρωπαϊκά ζητήματα και να είναι υπέρ των πολιτών, όχι εναντίον τους. Γι' αυτό και προτείνονται κάποιες αλλαγές στο σχέδιο έκθεσης, ώστε να αποφύγουμε περί το διοικητικό άχθος, το οποίο θα δημιουργήσει απογοήτευση στους πολίτες. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ελέγχει το παραδεκτό ή όχι κάθε πρωτοβουλίας αφού έχουν συγκεντρωθεί 300.000 υπογραφές. Ναι, αλλά μετά πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι μπορούν να ξεκινήσουν, θα μαζέψουν 300.000 υπογραφές και μετά θα ξεκινήσει αυτή η οχι καθε πρωτοβουλία, αφου εχουν συγκεντρωθει 300000 υπογραφες ναι αλλα μετα πως θα εξηγησουμε στους πολιτες οτι μπορουν να ξεκινησουν θα μαζεψουν 300000 υπογραφες και μετα θα ξεκινησει αυτη η διαδικασια θεωρήσαμε ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο και θελήσαμε να το αλλάξουμε. Γιατί μετά τι, θα σταματήσει δηλαδή η συλλογή υπογραφών, θα επαληθεύσει το παραδεκτό τη πρωτοβουλία η Επιτροπή και μετά θα συνεχίσουν ε, οι υπογραφέ. Θα είναι Γι' αυτό θέλω όμω γίνεται πιο νωρί στη διαδικασία σκόπος η συγκέντρωση όλων αυτών των υπογραφών. Γι' αυτό θέλουμε όσο γίνεται πιο νωρί τη διαδικασία να ελέγχει το παραδεκτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωράει κανονικά η συγκέντρωση υπογραφών. Έπειτα, άντε και μαζεύτηκαν οι υπογραφές. Θα έχει περάσει τόσος χρόνος. Και μετά η Επιτροπή θέλουμε έτσι κι αλλιώς να συναντιέται με τους πολίτες και να γίνεται μία κρόαση με τους πολίτες, ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσουν το θέμα τους και το αίτημά τους. Και η Επιτροπή θα πρέπει να απαντάει με επιχειρήματα, με πλήρη επιχειρήματα, δηλαδή κάτι να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέρφους να μας πούνε πώς θα γίνει πιο φιλική προς τον πολίτη αυτή η πρωτοβουλία και πώς θα αποφύγουμε καταχρήσεις. Θέλω να ακούσω τις σκέψεις σας επίσης για το ρόλο που έχει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία της πρωτοβουλίας αυτής. Με τον πρόεδρο Κασίνη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια σημαντική συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ο κύριος Ρότε από τη Γερμανία έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση και μας έδωσε πολλές ιδέες την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν την πέμπτη το απόγευμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από εσά τι βαθμό διαφάνειας επιθυμείτε και πώς θα τον πετύχουμε. Και όπως πάντα, ό,τι προτάσεις έχετε, ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι τον συνάδελφο Λαμασούρ, ο οποίο όμως είναι σε ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, Προπολογισμών και δεν μπορεί να είναι, στέλνει όμω το χαιρετισμό του. Να ξέρετε ότι από κοινού συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε. Αυτά τα λούδια είναι για την Σίλβια, Ακριβώ γιατί είναι η μητέρα τη πρωτοβουλία αυτή, εκ μέρου όλων μα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ευγενική αυτή χειρονομία επίσης της Αντιπρόεδρου κυρίας Κορμάη. Ποιος θέλει να παρεύει πρώτος από τους δύο προσκεκλημένους. Ο κύριος Μέγερα. Κύριε Πρόεδρε. Sehr geehrten Damen und θα κάνω μερικές προκαταρκτικές ε, παρατηρήσεις και θα έρθω μετά ε, σε μια τοποθέτηση επί του εξαιρετικού εγγράφου της εισηγητρίας. Πρώτα, επιθυμώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι πολλοί των ε, προσώπων τότε που είχαν αγωνιστεί μαζί μου τότε στην διακυβερνητική συνέλευση υπέρ της πρωτοβουλία των πολιτών. Πρώτα-πρώτα η Σίλβια Ιβόν Κάουχμαν, αλλά και ο Αλάλα Μασούρ επανέρχεται ως εισηγητής. Επίσης θα θυμίσω τον Γκέραλτ Χέφνερ, ο οποίος στην συνέλευση ήταν παρόν ως εκπρόσωπος ε, μη κρατικής οργανώσεως και αξίωσε περισσότερη δημοκρατία. Οι ενδιαφερόμενοι θα θυμούνται ότι στην ε, συνταγματική συνέλευση η πρώτη πρόταση που είχε αποβάλει με λίγες υπογραφές απορρίφθηκε από το Προεδρείο τότε. Αυτό είχε γίνει την άνοιξη του 2003. Ο λόγος ήταν ότι στο Προεδρείο της ε, Συνταγματικής Συνελεύσεως είχαν την πλειοψηφία οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και είχαμε τότε κατανοήσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν ήδη πρόβλημα με τα κοινοβουλιά τους είναι λοιπόν πολύ λιγότερο ε, ευχαριστημένοι να βλέπουν και άλλα στοιχεία άμεσης δημοκρατίας να τους απειλούν εντός εισαγωγικών. Ε, μετά όμως πολλά από τα μέλη της συνελεύσεως αλλά και ε, μη κρατικών οργανώσεων συνέλεξαν υπογραφές, συνολικά παραπάνω από 70 υπογραφές και την τελευταία ημέρα η πρωτοβουλία των πολιτών περιλήφθηκε τελικά στο σχέδιο της ε, συνελεύσεως τότε και που έγινε τώρα βεβαίως συνθήκη της Λισαβόνας. Για το λόγο αυτό, πολλοί ακόμη ελπίζουν να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες τροποποίησεις στο σχέδιο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένουν την υποστήριξη των βουλευτών. Οι βουλευτές, βουλευτές ήταν εκείνοι οι οποίοι κατόρθωσαν να επιτύχουν την πρόοδο τότε και οι βουλευτές είναι αυτοί που θα δώσουν τώρα την απαραίτητη όθηση. Δεύτερο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με το ότι εγώ στην διατύπωση της ε, πρωτοβουλίας εκείνης είχα επιλέξει την ίδια διατύπωση όπως και για το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνεται τώρα στο άρθρο 225 της ε, συνθήκης περί τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για να καταστεί σαφές ότι οι πολίτες αμφωτέρων των φίλων έχουν παρόμοια βαρύτητα, συγκρίσιμη βαρύτητα δηλαδή με την άσκηση της πρωτοβουλίας τους, έχουν δηλαδή την ίδια αξία οι πρωτοβουλίες αυτές όπως μια πρωτοβουλία που θα προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα η πρωτοβουλία των πολιτών δεν είναι ένα είδος ε, μαζικής αναφοράς η οποία απευθύνεται στο Κοινοβούλιο είναι μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται και που έχει παρόμοια βαρύτητα με αυτήν του Κοινοβουλίου και που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτη παρατήρηση. Όσο λιγότερο δεσμευτική είναι μια πρωτοβουλία, τόσο πιο γενναιόδωρα μπορεί να είναι κανείς σχετικά με τις προϋποθέσεις της. Αυτό ε, δεν έχει, αυτό έχει παραγνωριστεί νομίζω στο σχέδιο, διότι έχει επιβαρυνθεί με πολύ υπερβολική ε, γραφειοκρατία και ρυθμίσεις που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν νόημα σε μια μη δεσμευτική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα ότι στις υπογραφές πρέπει να δίνονται και ε, αριθμοί, προσωπικός αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων για παράδειγμα ή τέτοια πράγματα. Αυτό στο επίπεδο του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να είναι επιθυμητό, δηλαδή τέτοιου είδου υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτά ίσω να τα ορίσουν οι χώρε μέλη. Τελευταία μου παρατήρηση θα αναφέρεται στο ότι η πρωτοβουλία αυτή πολιτών έχει μια συγκεκριμένη έννοια. Να δημιουργηθεί δηλαδή στην ουσία μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, μια συζήτηση διαμεθοριακή. Οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα ε, να θέτουν θέματα, να φτιάχνουν δηλαδή όπως τα λέγαμε σε ε, μετάφραση από τις αγγλοσαξονικές γλώσσες, μια ατζέντα κοινή ευρωπαϊκή που να προωθούν θέματα δηλαδή και να μπορούν να προωθούν ε, τέτοια θέματα. Τώρα, δεν κατανοώ πως ορισμένοι, πολύ μάλλον, θεωρούν ότι στα θέματα των πρωτοβουλίων των πολιτών θα υπάρχουν δίθεν ορισμένα ταμπού. Δηλαδή κυρίως το ταμπού ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν οι πρωτοβουλίες αυτές με τροποποιήσεις ε, της συνθήκης, δηλαδή με συνταγματικό δίκαιο. Α υποθέσουμε ότι προβάλλει μια αξίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου απέναντι στην Κομισιόν να τροποποιήσει τι συνθήκε. Η Κομισιόν τότε ποτέ δεν θα πει Α, προσέξτε το θέμα αυτό είναι ταμπού. Γιατί στο 225 άρθρο σα προβλέπετε ότι μπορείτε να ασχολείστε μόνο με την εφαρμογή των συνθήκων. Το ίδιο όμως ε, γράφει και στο άρθρο 11 για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Όμως υπάρχει και το άρθρο 48 το οποίο προβλέπει τροποποίηση των συνθήκων μέσα σε μια τακτική διαδικασία. Μια δημοκρατία είναι ζωντανή μόνον εφόσον μεταρρυθμίζεται, ανανεώνεται γιατί λοιπόν οι πολίτες να μην έχουν ούτε καν την δυνατότητα να αρχίσουν μια συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανάγκη μεταρρύθμισης της συνθήκης. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ταμπού πρέπει να πέσει. Εφόσον μια πρωτοβουλία αναφέρεται σε τροποποίηση της συνθήκης, ασφαλώς βέβαια θα πρέπει ο καθένας, ή μάλλον η καθεμία από τις 27 χώρες μέλη να συμφωνήσουν. Άρα Ας μην γεννηθεί η ψευδέστηση ότι δήθεν οι πολίτες μπορούν να επιτύχουν μέσω της πρωτοβουλίας μια τροπή των συνθήκων. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μπορούν να θέσουν το θέμα υποσυζήτηση. Τώρα, για τα επιμέρους θέματα του εγγράφου εργασίας. που εξήτασα υπό το πρίσμα του τι θα πρέπει να συζητηθεί ακόμα. Τώρα, πρώτα το 3 που αναφέρεται στην ίδρυση μιας Επιτροπής Πολιτών από ένα τέταρτο των χωρών και μελή τουλάχιστον. Εγώ θεωρώ ότι πάλι πρόκειται εδώ για ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην είναι παράλογο να δημιουργηθεί ένας τέτοιος συνομιλητής, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να, είναι, πρέπει να προκαλούνται δυσκολίες στην διακρατική συνεργασία των πολιτών γιατί έτσι δίνεται η εντύπωση ότι μόνο οργανωμένα συνδικάτα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τι πρωτοβουλίε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή Πολιτών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύσταση, δεν θα πρέπει όμω να είναι υποχρεωτική. Τώρα, στο 5.1. Το ερώτημα δηλαδή που επιθυμούν να απαντηθεί οι εισηγητές Εάν δηλαδή η πρωτοβουλία θα πρέπει να συνδυάζει προσπάθειές της με εκλεγμένους ε, βουλευτές. Εδώ θεωρώ ότι είναι μια συμπερίληψη στοιχείου αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που δεν αρμόζει εδώ στην ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να εξαρτάται η ε, πορεία της πρωτοβουλία των πολιτών από το αν θα συμμετάσχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι όχι τρίτο. Το 5, 2. Μια κατάθεση ασφαλείας, δηλαδή πρόκειται εδώ για κάτι απολύτως απαράδεκτο. Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν οικονομικούς πόρους δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν ε, κάποια πρωτοβουλία. Άρα εδώ πρέπει να διαγραφεί χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Για το 8... Για την υποστήριξη δηλαδή των ε, πρωτοβουλειών θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητα διαφάνεια. Όσοι υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία πρέπει να είναι γνωστοί. Και το 9 τώρα, το οποίο ανέφερε ήδη η εισηγήτρια, αυτή η ατυχή ιδέα να συζητείτε το παραδεκτό μόνο αφήσει έχουν συγκεντρωθεί 100.000 ή 300.000 υπογραφές. Κατ' επανάληψη σε διάφορες ακροάσεις αλλά και στην προηγούμενη, εδώ, ε, και στην προηγούμενη ε, κοινοβουλευτική θητεία εδώ εγώ είχα ζητήσει να υπάρχει μονάχα μία εξέταση του παραδεκτού που θα πρέπει να γίνεται πριν από την καταχώρηση της πρωτοβουλία και θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν θα έχουν ε, συλλεχθεί 5, άντε το πολύ 10.000 υπογραφές. Για να μην θεωρούν οι πολίτες, να μην θεωρήσουν οι πολίτες ότι τους ε, ε, κοροϊδεύει κανείς όταν θα έχουν ήδη συγκεντρώσει 300.000 υπογραφές και θα τους πούνε μετά ότι είναι, ότι είναι μη παραδεκτή αυτή η ε, πρωτοβουλία. Και τώρα ε, αυτό το άλλο, το Συμβούλιο των Σοφών που υποτίθεται ότι θα απαλλάξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εξέταση του παραδεκτού. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι προβληματικό ως ιδέα, διότι η απορριπτική απόφαση κατά μιας πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αυτό, σύμφωνα με τη συνθήκη, μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αυτό το Συμβούλιο Σοφών θα είχε νόημα μόνο εάν είναι και καταληκτική η απόφασή τους. Γιατί τότε υπάρχει δυνατότητα να προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν πει δηλαδή το Συμβούλιο των Σοφών μάλιστα είναι παραδεκτό, τότε οκ, okay, να μην ασχοληθεί περαιτέρω η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε έχει κάποιο νόημα η απόφαση του Συμβουλίου των Σοφών και όχι να έρχεται υποχρεωτικά να μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 14.2 τώρα, εκεί, εδώ θέλω να τονίσω και πάλι την ε, σύμφωνη γνώμη μου για το ότι η τελική απόφαση στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να υποβάλλεται στην εξέταση από το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι πολίτες να μην έχουν την εντύπωση ότι για λόγους πολιτικούς ή κομματικούς εν τέλει απορρίπτεται η πρωτοβουλία τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δικαστική εξέταση εφόσον έχει ληφθεί απόφαση αρνητική κατά της πρωτοβουλίας. 19. Για την συλλογή των υπογραφών προβλέπεται περίοδος 12 μηνών αρχομένη από τις καταχωρήσεις. Εγώ νομίζω να ληφθεί εδώ υπόψη το ελβετικό παράδειγμα όπου είναι πολύ μικρότερα τα νούμερα και ωστόσο οι εμπειρίες που έχουν εκεί είναι πολύ θετικές με 18 μήνες. Ας μην λοιπόν σε 18 μήνες και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Τώρα 21 παράγραφος όπου προβλέπεται ακρόαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό είναι αυτονόητο. Λόγω του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, που από 1η Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους ισχύει δεσμευτικά. Έχω κάνει σχετικό σχόλιο στον εκδοτικό οίκο νόμος και μπορείτε να το διαβάσετε εκεί. Εδώ προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα και σε απόφαση χωρίς καμία καθυστέρηση οι πολίτες, αλλά και όταν υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα πρέπει η ακρόαση να είναι δημοσία. Εγώ παρακαλώ λοιπόν εδώ να μην γράψετε απλώς ακρόαση, αλλά δημόσια ακρόαση. Και επίσης προκύπτει από το 41, το 41, η καλή διαχείριση η χρηστή διοίκηση και επίσης η απόφαση να ε, ανακοινώνεται, να εκδίδεται ε, στην γλώσσα των πολιτών ή τουλάχιστον στις γλώσσες των 7 χωρών από τις οποίες προέρχονται υπογραφές. 9 γλώσσες είναι υπερβολικές, 7 χώρες, 7 γλώσσες, εφόσον είναι κάθε μια ξεχωριστή, που θα απευθύνεται ε, στη διοίκηση. Αυτό είναι και το νόημα της χρηστή διοίκηση ε, σύμφωνα με το χάρτη των δικαιωμάτων. Και τελευταία παρατήρηση, η ιδέα ότι θα εκδηθεί ένα εγχειρίδιο χρήστου για την πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά καλό. Δείχνουμε τον τρόπο αυτό ότι ναι, μα ενδιαφέρει η πρωτοβουλία των πολιτών και θέλουμε να σα βοηθήσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε διαρκώς γραφειοκρατικά εμπόδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, ήσασταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και λακωνικό. Θα ανταλάβουμε υπόψη όλα όσα μα είπατε. Και τώρα παρακαλώ το λόγο στην δόκτωρα Σίλβα Ιβον Κάουφμαν. σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς ιδίως κύριε Πρόεδρε αλλά και τους δύο ζητητές για την πρόσκληση να προσέλθω σήμερα ενώπιόν σας. Θα μπορείτε να φανταστείτε ότι για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή η παρουσία μου σήμερα εδώ. Μετά από τόσα χρόνια που έχω αγωνιστεί υπέρ του θέματος αυτού είναι πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη ικανοποίηση που βλέπω σήμερα ότι οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτέλους προχωρούν στην λήψη των απαραίτητων μέτρων για να δώσουν σάρκα και οστά στην ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Σας εύχομαι βεβαίως καλή επιτυχία στην προσπάθεια αυτή. Ελπίζω από την έκθεση αυτή να προκύψει ένας κανονισμός γιατί όλοι εργαστήκαμε υπέρ της ιδέας αυτής ώστε να προσφέρουμε κάτι στους πολίτες να αντιληφθούν οι πολίτες ότι, είναι, ότι το project της Ευρώπης είναι κάτι που τους αφορά και η, αυτή, η προσπάθεια αυτή να έχει γίνει από πλευράς μας. Σήμερα έχω υποβάλει ήδη ένα έγγραφο θα διανεμηθεί, ελπίζω και πιστεύω, μετά από την συζήτηση στους βουλευτές. Εγώ εξέτασα τα έγγραφα που ήταν διαθέσιμα, δηλαδή και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έγγραφο εργασίας που είναι πραγματικά εξαιρετικό των δύο συγητών, αλλά και τις γενικές κατευθύνσεις του Συμβουλίου του παρελθόντος Ιουνίου Αυτά τα έγγραφα δίνουν μια εικόνα του πού βρίσκεται και προς τα πού κινείται η συζήτηση και στα τρία θεσμικά όργανα. Θα συμφωνήσω απολύτως με τα όσα είπε ο καθηγητής Μάιερ, ότι δηλαδή το κεντρικό κριτήριο για την επεξεργασία του κανονισμού θα πρέπει να είναι για όλους ο εύχριστος χαρακτήρας του εργαλείου αυτού, το οποίο πρέπει να αποβεί ελκυστικό για τους πολίτες και πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευθεί η αδίποτε απογοήτευση από πλευρά πολιτών. Η υλοποίηση δηλαδή της των πρωτοβουλειών αυτών να είναι εύκολη. Έχοντας υπόψη τα τρία έγγραφα που ανέφερα πριν, θα αναπτύξω οχτώ ε, ζητήματα που όλα φωτίζονται από το φως αυτό, δηλαδή της ευχρηστίας... της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Από την σκοπιά μου, ο ελάχιστος αριθμός των κρατών όπου θα συλλέγονται οι υπογραφές θα πρέπει σαφώς να είναι κάτω του ενός τρίτου του αριθμού των χωρών μελών. Εάν εξετάσει κανείς την θεμελίωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει δηλαδή την ενισχυμένη συνεργασία. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι πιστικό το επιχείρημα αυτό, διότι το, ο μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας είναι πολύ εξειδικευμένος που έχει σκοπό να επιτρέψει σε έναν αριθμό χωρών να προχωρήσουν μόνο εφόσον δεν διαγράφεται πλειοψηφία μέσα στο Συμβούλιο Υπουργών. Εδώ όμως μιλούμε για διαδικασίες νομοθετικές, για το, την ανάλυση του πρώτου βήματο, μια πρώτη πρωτοβουλία για το ξεκίνημα μιας νομοθετικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι ακόμα και το 1 τέταρτο είναι υπερβολικό όταν μιλούμε για το ξεκίνημα μιας διαδικασίας νομοθετικής θα μπορούν να είναι 6, 5, ίσως και 4 χώρες. Εφόσον Πολίτε από τέσσερις χώρες δείχνουν ενδιαφέρον, σημαίνει ότι ήδη το θέμα αυτό είναι σημαντικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο που το έθιξε επίση ο κύριος Μάιερ, το υποστηρίζω και εγώ, η εξέταση του παραδεκτού της ε, πρωτοβουλία πολιτών προτείνει η Επιτροπή να γίνεται είτε άμα τη συλλογή των 300.000 υπογραφών ή των 100.000 υπογραφών σύμφωνα με το Συμβούλιο. 300.000 ε, η Κομισιόν, 100.000 το Συμβούλιο. 300 η Εγώ θεωρώ ότι η εξέταση του παραδεκτού θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην βάση σαφώς ορισμένων νομικών κριτηρίων. Δηλαδή, πρωτοβουλίες των πολιτών θα πρέπει να απορρίπτονται μόνον εφόσον παραβιάζουν τις αρχές του άρθρου 2 ή τις αρχές του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ή εκπίπτουν των πλαισίων των ε, συνθήκων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ε, διαγράψει κανείς και το άρθρο 4 παράγραφος 3 που ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να απορρίπτονται καταχρηστικές ή προφανώς άσκοπες ε, πρωτοβουλίες ε, πολιτών. Η εξέταση του παραδεκτού θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται έγκαιρα, σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Συμφωνώ με τους ηγητές. Άμα τη συλλογή 5.000 υπογραφών. Αν ληφθεί αυτό ως κριτήριο, δεν χρειάζεται να ληφθεί, δεν χρειάζεται να ιδρυθεί ε, και αυτή η επιταμελής επιτροπή που βρίσκω ότι είναι κάπως γραφειοκρατική. Ίσως κάποιες μεγάλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για παράδειγμα μεγάλα συνδικάτα, μπορούν να έχουν ε, την πολυτέλεια αυτή, αλλά για τους ε, πολίτες ατομικά, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι υποχρεωμένοι εξ αρχής να ιδρύουν επιτροπή Επτά μελών. Τώρα, για την ε, Επιτροπή ή το Συμβούλιο των Σοφών ε, τοποθετούμε στο εγγραφό μου. Ε, θεωρώ ότι δεν είναι σκόπιμο. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα περαιτέρω περιττό κόλλημα. Διότι και οι ίδιοι οι συγκητές γράφουν στο έγγραφο εργασία τους ότι εν τέλει ή το θέλει κανεί είτε όχι, την απόφαση τη λαμβάνει η Κομισιόν, η οποία φέρει και την ευθύνη και δεν θα πρέπει να απαλλάσσετε τις ευθύνες αυτής με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν. Όπως είπε και ο Μάιερ προηγουμένως, το θέμα τίθεται εδώ και ενδεχομένως στα πλαίσια προσφυγής επί ακυρώσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εξέταση του παραδεκτού και καταχώρηση στην ουσία πρέπει να είναι το ίδιο βήμα. Μόνο παραδεκτές πρωτοβουλίες πολιτών θα μπορούν να καταχωρίζονται και μάλιστα από το παραδεκτό μέχρι την καταχώρηση υπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος δύο μηνών διότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν προσφυγές για ακύρωση ενδεχομένω από μια χώρα μέλο κατά τι αποφάσει της Κομισιόν. Τέταρτον, το περιθώριο των 12 μηνών για την συλλογή των υπογραφών είναι πολύ περιορισμένος, πολύ περιορισμένο ο χρόνος αυτός. Ε, μιλούμε για μια Ευρώπη με πλήθος ε, χωρών μελών, με πλήθος γλωσσών, θα πρέπει να ε, προτιμήσουμε 18 μήνες. Πέμπτο, πρόταση της Επιτροπής υπερβολικά γραφειοκρατική, αυτή δηλαδή που προβλέπει να αναφέρονται στις συλλογές των υπογραφών αριθμοί προσωπικών ταυτοτήτων, αριθμοί ε, κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ. Αυτό είναι αποτρεπτικό για τους πολίτες. Όποιος έχει συλλέξει υπογραφές ε, στον δρόμο και προσπαθεί να κερδίσει το ενδιαφέρον των πολιτών, μπορεί να φανταστεί ότι ο κάθε πολίτης θα ε, τρομάξει και θα ε, διστάσει. Ε, θα πει, μα πώς, γιατί θέλετε την αριθμό ταυτότητάς μου. Έκτο, η συγκήτρια το είπε επίση στην αρχή και το υποστηρίζουμε και εμείς, οι οργανώτριες και οργανωτές μιας επιτυχημένης πρωτοβουλίας πολιτών, εφόσον δηλαδή έχουν συλλεχθεί όντω ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκτούν δικαίωμα ακροάσεως από την Κομισιόν και μάλιστα η ακρόαση αυτή να είναι δημοσία διότι θεωρώ ότι η αποκατάσταση αυτή διαλόγου μεταξύ πολιτών και Κομισιόν που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα πρωτοβουλίας και από την πρωτοβουλία των πολιτών αυτών θα ξεκινήσει μια νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν, χρειάζεται οπωσδήποτε τέτοια επικοινωνία διότι με ένα απλό μόνο στη βάση ενός εγγράφου το οποίο, στο οποίο θα αναγράφονται οι στόχοι της ε, πρωτοβουλία πολιτών δεν μπορεί να γίνει η προσπάθεια αυτή. Θα δείτε στο εγγραφό μου ότι προτείνω επίσης να σκεφτεί η Κομισιόν αν ίσως επιθυμεί να ιδρύσει ένα γραφείο πρωτοβουλίων πολιτών θα προέκυπτε αυτό και από το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπου οι οργανώτριες και οι οργανωτές να μπορούν να λαμβάνουν και πληροφορίες από την Κομισιόν. Για παράδειγμα, εάν για το θέμα που θέλουν να αρχίσουν μια πρωτοβουλία υπάρχει ήδη ίσως μια ε, έναρξη νομοθετικής πρωτοβουλίας ή αν υπάρχει κάποια, αν διαγράφεται κάποια άλλη ε, πρωτοβουλία πολιτών. Άρα εκεί θα προσφέρει υπηρεσίες η Κομισιόν ε, στους πολίτες. Έβδομο, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εάν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως άμεσα εκλεγμένο όργανο εκπροσώπηση των πολιτών να λάβει τη δέσμευση και αυτό να ε, ακροαστεί δημοσία των ε, οργανωτών. Να προβάλλει δηλαδή με τη σειρά του και αυτό την πρωτοβουλία των πολιτών. Και να λάβει θέση από αυτής. Το 8ο, ή στα τρία έγγραφα θεωρείτε ότι η στα τρια εγγραφα θεωρείται οτι η το ελάχιστο όριο ηλικία για τη συμμετοχή σε πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι η ηλικία που επιτρέπει το δικαίωμα του εκλέγην. Για μένα αυτό είναι σαφές. Στις περισσότερες χώρες μέλη ισχύουν τα 18 έτη της ηλικίας. Μόνο σε μία χώρα, δηλαδή στην Αυστρία, θα, είχαμε την, ε, θα υπήρχε η δυνατότητα να αρχίζουν ε, να μπορούν οι πολίτες να ξεκινήσουν πρωτοβουλία πολιτών για από τα 16 τους χρόνια. Οι ε, οσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι αντίθετος με τις αρχές μας. Νομίζω λοιπόν ότι υπό το φως αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και πάλι αν ίσως είναι σωστό να ισχύσει σε όλη την Ένωση ένα όριο ηλικίας και αυτό να κατέβει στο ελάχιστο, δηλαδή στα 16 χρόνια. Άλλωστε και το δικαίωμα αναφοράς δεν περιορίζεται. Γιατί άραγε να περιοριστεί εδώ στην πρωτοβουλία πολιτών. Εν τέλει, έρχομαι σε κάτι που είπε ο καθηγητής Μέιερ ήδη στην αρχή της ομιλίας του, τότε με τη δική μου έκθεση είχαμε συζητήσει διαμακρών σχετικά με το εάν η διατύπωση του άρθρου 11.4 σημαίνει επίσης ότι πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει ενδεχομένως να είναι παραδεκτή και για τροποποίηση της συνθήκης. Εν τέλει, ε, μεγάλη πλειοψηφία είχε ταχθεί κατά. Και πολιτικά ωστόσο νομίζω δεν μπορούν να αγνοήσουν ε, τα θεσμικά όργανα το ενδεχόμενο οι πολίτες να ζητούν μια τροποποίηση της συνθήκης. Και εφόσον αυτή νομικά απευθύνεται στην Κομισιόν, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θέλω τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί εάν ίσως το ίδιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει πρωτοβουλίες πολιτών που θα απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον τίθεται θέματα θεσμικά, συνταγματικά, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το ίδιο το δικαίωμα να υποβάλει σχέδια τροποποίησεων της συνθήκης και εδώ, όντας και άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα έχει το δικαίωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που να δέχεται πρωτοβουλίες ε, των ε, πολιτών. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε και τα αιτήματα πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η τελευταία πλέον τροποποίηση των αρχικών συνθήκων. Θα ήταν δυνατόν λοιπόν να σκεφτεί κανεί ότι μπορεί να γίνουν προτάσει με, με ένα εκατομμύριο υπογραφέ. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι κύριε Πρόεδρε και εύχομαι καλή επιτυχία στην περαιτέρω πορεία τη ε, πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κάφμαν. Βουλευτά Κάφμαν, γιατί ξανήρθατε εδώ στη θέση σας που είχατε στο Ευρωκοινοβόλιο, στην ίδια Επιτροπή, προσωρινά τουλάχιστον. Και αρχίζει η συζήτηση. Ποιος θέλει να μιλήσει. Scholz. Ähm, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τους δύο ειδικούς, οι οποίοι επί χρόνια εργάζονται επί του θέματος είτε στη Συνταγματική Συνέλευση είτε και στην Ευρωβουλή είτε και εκτός συμφωνώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις απόψεις τους νομίζω ότι και οι ακροάσεις που έχουμε διεξαγάγει στις διάφορες ε, πολιτικές ομάδες της θύμισε και η Αγκουρμάη ή και πολλές συζητήσεις που έχουμε διεξαγάγει στις επιτροπές έχουν επιτρέψει μια πραγματικά λεπτομερή εξέταση του αντικειμένου και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περάσουμε ως πολιτικό μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τους πολίτες. Πρόκειται για μηχανισμό, για εργαλείο που θα επιτρέπει την συμμετοχή στο δημοκρατικό γίγνεσθε των πολιτών. Και η υψίστη επιταγή θα πρέπει να είναι αυτή. Μιλούμε τώρα βεβαίω για τα επιμέρους, παραγράφους, υποπαραγράφους κτλ. Αλλά νομίζω ότι και εξ ονόματο της πολιτικής μου ομάδας μπορώ να πω ότι όπου στην ομάδα μου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δεν το αποσιωπώ αυτό, υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις, αλλά να εξευρεθεί μια ρύθμιση η οποία να ε, κατεβάζει το κατόφλι έτσι ώστε να επανέλθουν στην εργοπολιτική ζωή οι πολίτες αυτό θα πρέπει να είναι ε, αυτό που θα πρέπει να μας κινεί. Και γι' αυτό συμφωνήσω με τους κυρίους Κάφμαν και Μέιερ. Τώρα, δύο-τρεις μικρέ ερωτήσεις. Τίθεται το ερώτημα τι είναι επί της ουσίας παραδεκτό. Δηλαδή θα είναι και πρωτοβουλίες πολιτών που ε, ενδέχεται να αποζητούν την τροποποίηση των πραγματικότητων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους αγγίζουν καθημερινά και έντονα. Ε, νομίζω ότι και εκεί πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη τους πολίτες. Οι, οι πολίτες δεν θα θέλουν να καταστρέψουν την Ένωση, αλλά ασκούν κριτική πάνω στη μια ή στην άλλη εξέλιξη. Εκεί λοιπόν το παραδεκτό πρέπει να αναγνωρίζεται από άψη ε, πολιτική για να ασχοληθεί δηλαδή ένα θεσμικό όργανο. και ω ενάσμα για μια νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν. Ή, επίσης, κάτι που μου φαίνεται ιδιαίτερα επιθυμητό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιφυλάξει σε αυτόν το δικαίωμα μέσω του κανονισμού του να πει ότι ναι, παίρνουμε σοβαρά υπόψη μια τέτοια πρωτοβουλία ακόμα και αν έχει 900.000 υπογραφές. Την λαμβάνουμε τότε υπόψη μέσα στην πρωτοβουλία αυτή και εγκύπτουμε εμείς σε αυτήν. Ε, δεύτερο σχόλιο, η ηλικία. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να ισχύσουν τα 16 χρόνια. Το έδειξε και η συνάντηση με τις Εθνικές Βουλές. Η ιδέα αυτή είναι πολύ διαδεδομένη. Και εδώ νομίζω ότι αυτό είναι μια έμεση πρόσκληση προς τους ε, πολίτες να ασχοληθούν με τα κοινά. Και το συζητήσαμε και με τον ΤΑΦ που κάνει σχετική έκθεση για την ε, τροποποίηση του εκλογικού ε, συστήματος. Εμείς θέλουμε την δημοκρατική διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε την συμμετοχή των νέων πολιτών και γι' αυτό νομίζω ότι τα 16 χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Εν τέλει, η εξέταση του παραδεκτού. Και αυτή θα πρέπει να αποτελεί ένα χαμηλό κατόφλι, εύκολο να το διαβούν. Στην αρχή, λοιπόν, με πολύ μικρό αριθμό, οι δεμοί στην ουσία θα προκαλέσουμε πάλι απογοήτευση των πολιτών. Εγώ λέω 3.000 υπογραφές. Καλά, έστω 5.000 υπογραφές, αλλά από το δυνατόν λιγότερες χώρες. Κατά τα άλλα, ε, εύχομαι και εγώ στους εισηγητές θάρρος και καλή επιτυχία ε, στην ε, περαιτέρω πορεία της εκθέσεως. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι εδώ τακτικό μέλος στην Επιτροπή αυτή. Με ενδιαφέρει όμως πολύ το θέμα. Είμαι Ολλανδός, ο οποίος εκλέγεται στο Βέλγιο. Και συμφωνώ και εγώ αν υπάρχουν υποψηφιότητε από ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ολλανδία διαπίστωσα όταν συζητούσαμε για το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ότι υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες οι πολίτες να εκφραστούν. Και όταν εκφράζονται, ε, τελικά εκφράζονται από θυμό και είναι αρνητικοί. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών που υπάρχει στη Γερμανία εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι πολύ θετική και συμφωνώ εδώ με τον διπλανό μου, παρόλο που είναι από άλλη πολιτική ομάδα, ε, με αυτά που είπε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συζητητές και τον κύριο Μάγερ και την κυρία Κάφμεν ε, για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση αυτή. Σε ένα θέμα θέλω να αναφερθώ εγώ και ίσως να πιστήσω έτσι την ε, προσοχή της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής. Έχει να κάνει με την στήριξη, με τις υπογραφές και την επαλήθευση των υπογραφών αυτών. Τι στοιχεία πρέπει να δίνει κανείς. Λέμε αριθμό ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης ή διαβατηρίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς πολίτες. Εγώ γνωρίζω πολλές χώρες όπου οι πολίτες αρνούνται να δώσουν τέτοια στοιχεία, γιατί πίσω από τα στοιχεία αυτά υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμος. Πίσω από τον αριθμό ακριβώς ταυτότητας υπάρχει μια ολόκληρη ταυτότητα. Και η γενιά που πέρασε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ δεν θέλει, αρνείται, ε, αντιστέκεται έτσι κι αλλιώς να συμπληρώσει ηλεκτρονικά ένα έγγραφο. Ακριβώ γιατί φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν καταχρήσει κλπ. ή να μάθουν άλλοι πράγματα που γίνανε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία πολιτών ελπίζω η Επιτροπή αυτή να στηρίξει μια πρωτοβουλία με την οποία να ζητάει να μην απαιτείται αριθμό ταυτότητα διαβατηρίου κοινωνική ασφάλιση κτλ. Να βρεθεί ένα άλλο τρόπο επαλήθευση και να μην είναι αναγκαίο. Στο κάτω-κάτω δεν έχουν σε όλε τι χώρε όλοι οι πολίτε έναν αριθμό διαβατηρίου. Και άρα δεν μπορεί να εντοπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες να προστατεύουμε τον ιδιωτικό βίο των πολιτών γιατί αλλιώς δημιουργείται ένα εμπόδιο για τους πολίτες και οι πολίτες δεν θα είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες, κάτι το οποίο θα οδηγήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να θυμώσουν ακόμα περισσότερο σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το είδαμε αυτό και στην Ολλανδία στο κάτω-κάτω τότε που είχαμε το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τώρα, ο εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών, ο κύριος Έπνερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. και τους δύο ειδικού που είχαν συμβάλει σημαντικά και τότε στη Σταγματική συνέλευση και γι' αυτό και είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα σκεπτόμουν να ρωτήσω σχετικά με το νόημα της πρωτοβουλίας αυτής. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως σχολιαστές ή εν πάση περιπτώσει εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά. Σημαντικό λοιπόν που τους έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Με την ευκαιρία αυτή έχω ορισμένε ερωτήσεις να τους υποβάλω, αλλά θέλω να εκφράσω και τη λύπη μου διότι αντίθετα με αυτά που ανέμενα δεν έχω λάβει όλα τα έγγραφα. Για παράδειγμα δεν έχω λάβει το έγγραφο εργασίας των δύο εισηγητών της Επιτροπής Αναφορών με την οποία συνεργαζόμαστε. Το βρίσκω κρίμα λοιπόν ότι στη διαθεσή μας είχαμε μόνο ένα μέρος των εγγράφων. Καλά, αρκούμε σε αυτό το σχόλιο. Αλλά αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα ερωτήματα που δεν έχουν τεθεί. Μία πρώτη ερώτηση σχετικά με την διαφάνεια του οικονομικού υπόβαθρου των πρωτοβουλειών. Δηλαδή η ιδέα ότι οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να προβούν σε κάποια κατάθεση, σε κάποια παρακαταθήκη, αυτή δεν θα ισχύσει, αλλά υπάρχει ωστόσο η ιδέα, η κοινή γνώμη, να πληροφορείται ποιος χρηματοδοτεί εν τέλει την πρωτοβουλία αυτή. Εδώ μας ενδιαφέρει ιδίω το ερώτημα πότε, σε ποιο χρονικό σημείο δηλαδή, μπορεί κανείς να απαιτήσει να γίνει γνωστή η πληροφορία αυτή. Δεύτερο, το ερώτημα της εξέτασης του παραδεκτού. Θα ρωτήσω τον κύριο Μάιο ή και τους δύο που εκφράστηκαν επιφυλακτικοί για το θέμα των 7. Αλλά έχει σχέση τώρα και με τις 300.000. Η Κομισιόν φοβείται ότι μπορεί να υπάρξει πλημμυρίδα μη σοβαρών πρωτοβουλειών που θα καλύψουν κάποιες που ενδεχομένω είναι σοβαρές. Γι' αυτό και πρότεινε η Κομισιόν πρώτα 300.000 υπογραφές και μετά εξέταση του παραδεκτού. Εδώ οι συγητές είναι όλοι σύμφωνοι ότι η πρόταση αυτή είναι αδύνατον να εφαρμοστεί. Η πρόταση των εισηγητών να ζητήσουν πρώτα 7 υπογραφές αλλά αυτό σημαίνει και ένα τεστ της σοβαρότητας. Δηλαδή δεν θα θεωρείται και το τελευταίο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που, λαμβάνει, που αποστέλει κανένας μέσα στα νεύρα του επειδή κάτι δεν του άρεσε να θεωρείται ως αρχή πρωτοβουλία. Τουλάχιστον έχουν συλλεχθεί 7 υπογραφές. Τώρα, για την επαλήθευση. Με ενδιαφέρει εδώ περισσότερο νομικά. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε. Μας ενδιαφέρει η ατομική ταυτοποίηση του κάθε υπογράφοντος. Εξάλλου, ο επιτετραμένος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Λέει ότι θα, θα παραβούμε την νομοθεσία αν το ζητήσουμε αυτό. Ή πρέπει απλώς να είναι δυνατόν να ε, διαπιστωθεί εάν Α υπάρχει, αν Α υπάρχει το πρόσωπο αυτό πραγματικά, Β έχει το δικαίωμα να υπογράφει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δε, ε, επίσης θα ήθελα να υπάρξει μια συμπλήρωση διότι προηγουμένως λέχθηκε ότι ενδεχομένως οι χώρες μέλη μπορούν να το ρυθμίσουν αυτό η καθεμιά με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, η ιδέα των εισηγητών είναι περισσότερο ότι μια διαφορετική μεταχείριση του θέματος από χωρών μελών δεν είναι σωστή. Διότι η ρύθμιση αυτή θα οδηγούσε εν τέλει σε ένα patchwork στην Ευρώπη, όπου αλλού θα ήταν εύκολο, αλλού θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει κανεί σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή, πανενωσιακή δηλαδή ρύθμιση, που θα λέει ότι ενδεχομένως πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, η εθνικότητα, ο τόπος διαμονής. Αυτά θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένα ότι και θα μπορεί λοιπόν με έλεγχο να διαπιστωθεί αν το πρόσωπο υπάρχει και αν, είναι, αν έχει το δικαίωμα να υπογράφει τέτοια πρωτοβουλία. Μία τελευταία ερώτηση. Έχει γίνει πρόταση οι πολίτες όταν καταθέτουν τέτοια πρωτοβουλία πολιτών να επικαλούνται και τη νομική βάση της πρωτοβουλίας τους. Εδώ εκφράζονται βέβαια από τους φοιτητές και σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με το ότι αυτό ενδέχεται να είναι υπερβολικό βάρος, υπερβολική επιβάρυνση. Γνωρίζουμε συχνά ότι το θέμα της νομικής βάσης πολύ συχνά είναι από τα πιο δύσκολα να επιληθούν σε ένα κανονισμό. Και εδώ, στις δικές μας συζητήσεις, εδώ λοιπόν τίθενται ερωτήματα από πλευρά συζητητών και θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να τοποθετηθείτε. Τελευταία μια παράκληση προς τον καθηγητή Μάιερ. Σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να είναι παραδεκτές πρωτοβουλίες οι οποίες ζητούν την περαιτέρω εξέλιξη των συνθήκων. Κύριε Μάιερ, σχολιάστε αυτό που είπε η κυρία Κάφμαν. Και τι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δικές μας ρυθμίσεις, ώστε να κινηθεί εκ παραλίλου αυτό που ε, διαμορφώνουμε εμείς εδώ και με το Κοινοβουλίο. Ευχαριστούμε κύριε Έφνερα. συνάφο Ετερμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ισπανικά. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένα σχόλια. Τις τελευταίες ε, μέρες είδαμε ότι έγιναν διάφορες συναντήσεις και σεμινάρια με θέμα την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Και σε όλες αυτές τις συναντήσεις υπόθηκε το ίδιο, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τους πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι μιλάμε εδώ πέρα για πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Είναι Πολύ σημαντικό λοιπόν να το συζητήσουμε και να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να φοβάται τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα σύμπτωμα. Σύμπτωμα που απορρέει από την πολιτική κρίση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν θέλω να είμαι βέβαια πολύ αρνητική, όμως για μένα η συζήτηση αυτή με βάζει σε πολλές σκέψεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρή και αξίζει τον κόπο να καθίσουμε και να σκεφτούμε κατά πόσο τελικά θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ή όχι. Αν πραγματικά θέλουμε να τους ακούσουμε, εντάξει τότε, ας προχωρήσουμε με την πρωτοβουλία αυτή των πολιτών. Αλλά αν αποφασίσουμε ότι τελικά δεν θέλουμε να τους ακούσουμε και η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών δεν είναι παρά μια πρόφαση, αν απλώς θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε απέναντι στους πολίτες, δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε. Εγώ φοβάμαι ότι ακριβώς προχωράμε με την πρωτοβουλία αυτή μόνο και μόνο για να βελτιώσουμε την εικόνα μας, το image μας. Αλλά τότε καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι η κρίση. Ας το σκεφτούμε αυτό, ας καθίσουμε να το σκεφτούμε σε βάθος και να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν τέτοιες πρωτοβουλίες και για να τροποποιούν τις συνθήκες και για να θέτουν γενικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες, με τις εντολές, με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους φοβόμαστε. Το επαναλαμβάνω αυτό. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε περιορισμούς πολλούς θα σας μιλήσω λιγάκι για τη συνεργασία που έχουμε στις, στη Βόρεια Ευρώπη. Δέκα χρόνια ήμουνα στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών και κάποια μέρα όταν οι βόρειες χώρες έγιναν ε, μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχασε βέβαια το βάρος του το Συμβούλιο αυτό. Πριν όμως από αυτό, το Συμβούλιο αυτό Βορείων Χωρών ήταν πολύ σημαντικό και ήταν κάτι σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της βέβαια. Η αγορά ήταν κοινή, ενιαία, πιο πολύ μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκείνο από το Βόρειο Συμβούλιο από ό,τι τώρα. Δεν χρειαζόμασταν διαβατήρια, ένα σωρό πράγματα. Ήδη μεταξύ μας στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών όλα αυτά είχαν καταργηθεί. Γινόντουσαν ε, προτάσεις και τα κοινοβούλια τις προθούσαν. Έτσι συνέχισε να λειτουργεί το Συμβούλιο Βορείων Χωρών. Υπήρξαν βέβαια διάφορες επικρίσεις, αλλά από την άλλη μεριά ο κόσμος το εκτιμούσε όλος ιδιαίτερος. Γιατί ο κόσμος ήθελε να πηγαίνει στο Συμβούλιο αυτό. Θυμάμαι τι λέγανε οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλαν ε, σαν τρελοί να αποτελούν μέρος του Συμβουλίου αυτού, γιατί μέσα σε αυτό το Συμβούλιο συμβαίναν πράγματα και δεν φοβόμασταν τους πολίτες. Η εμπειρία δικιά μου είναι ότι από τον κόσμο έρχονται καλές προτάσεις. Όπως έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Κοινοβούλιο. Εννοείται ότι και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνουν και αυτοί κακές προτάσεις. Οπότε επαναλαμβάνω, μην φοβόμαστε τους πολίτες. πρέπει να έχουμε μια πρωτοβουλία εύχρηστη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Η πρωτοβουλία αυτή όταν αρχίσει να λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο, στις διάφορες χώρες μέλη, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, πώς θα επαληθεύονται οι υπογραφές, πώς θα λειτουργήσει επιτόπου Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο εδώ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όμως τις εμπειρίες που έχουμε από τα κράτη-μέλη και από αυτές εμείς να αντιγράψουμε την καλύτερη πρακτική. Οπότε σας είπα, να αποφασίσουμε θέλουμε πραγματικά μια πρωτοβουλία πολιτών που να αξίζει το όνομά της ή όχι. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα δανέζικα. Συμφωνώ με πολλά από τα κριτικά σχόλια τα οποία ακούσαμε. Όσο με τα προσκόμματα που υπάρχουν προκειμένου να εγκριθεί αυτή η κίνηση. Αλλά πέρα από το, τα τυπικά εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά το αποδεκτό ή όχι, Υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά τις συγκεκριμένες αντιρρήσεις της Κομισιόν, όπως εκφράζονται στο άρθρο 4 υπό παράγραφο 3 και 4, που μεταξύ άλλων προτείνει μια αξιολόγηση σχετικά με το πόσο λογική είναι η πρόταση. Αν πάρουμε 100 άτομα που συζητάνε για το πόσο λογικό είναι κάτι, πόσο ενοχλητικό είναι, σίγουρα θα έχουμε 100 διαφορετικές εκτιμήσεις. Γι' αυτό αυτό το άρθρο μάλλον θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες όσον αφορά την αξιολόγηση. Και αυτό νομίζω δεν βοηθάει κανένα. Είναι περίεργο. Τότε στην παράγραφο 4 αποφασίζεται ότι μικρά τμήματα της συνθήκης θα αφαιρεθούν προκειμένου να αποτελέσουν κριτήριο νομιμότητας που σημαίνει ότι το άρθρο 6 της συνθήκης περιέχει ορισμένα στοιχεία και γίνεται αναφορά σε αξίες. Τι γίνεται όμως με την αρχή της επικουρικότητας, της αναλογικότητας. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση που να λέει ότι θα πρέπει να το δούμε και κάτω από αυτό το πρίσμα. Νομίζω ο λόγος είναι διότι θα υπάρξει ενδεχομένως η δυνατότητα για υποκειμενικούς λόγους να σταματήσει μια πρωτοβουλία μια επιθυμητή. Αν είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί κανείς να τη σταματήσει πριν καν φτάσει στο 1 εκατομμύριο υπογραφές που απαιτούνται. Κανονικά θα έπρεπε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, να πούμε ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τη βάση της συνθήκης. Δεν μπορούμε να πάρουμε μόνο ένα τμήμα της συνθήκης με βάση αυτό να κρίνουμε. Θα πρέπει να είναι το σύνολο της συνθήκης, όχι μόνο το άρθρο 6 των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. Άρα, όλη η συζήτηση αυτή για το παραδεκτό ή όχι είναι ενδιαφέρουσα μεν, αλλά δίνει τη δυνατότητα, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, σε ομάδες πολιτών να αισθάνονται ακόμη περισσότερο στο περιθώριο της Ένωσης. Γιατί ποιος θα πει ναι ή όχι σε αυτό. Εμείς έχουμε ένα εκατομμύριο πολίτες που ξεκινάνε μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να ακολουθήσει την κανονική νομοθετική διαδικασία, κομισιόν, συμβούλιο, κοινοβούλιο. Εμείς, όπως κάνουμε οποιαδήποτε άλλη πρόταση της κομισιόν, θα πούμε το ναι ή το όχι. Γιατί μην έχει και ο πληθυσμό, οι πολίτες το ίδιο δικαίωμα. Και γιατί εμείς ως πολιτικοί να μπορούμε να πούμε όχι σε κάτι που δεν θεωρούμε σωστό. Αν ένα εκατομμύριο πολίτες στην Ευρώπη. Προωθούν μια λογική πρόταση. Νομίζω έχουν το ίδιο δικαίωμα όπως και εμείς εδώ. Δεν θα έπρεπε μια ομάδα υπαλλήλων της Ένωσης να αποφασίζουν κάτι είναι παραδεκτό ή όχι. Οι πολιτικοί θα πρέπει να το κάνουν αυτό. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι στο ύψος των υποχρεώσεών τους έναντι του εκλογικού του σώματος. Και η διατύπωση αυτή που περιορίζει το τι μπορούν να υποβάλουν ένα εκατομμύριο πολίτες ως πρωτοβουλία είναι απαράδεκτη. Και αν αφαιρέσουμε, αν πάρουμε μόνο ένα τμήμα της συνθήκης και μόνο, μόνο αυτό το τμήμα έχει σημασία, αυτό δεν είναι σωστό. Φοβόμαστε όχι μόνο του πολίτε φοβόμαστε και εμά του ίδιου. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μα ότι θα είμαστε σε θέση να πούμε ναι ή όχι σε μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ σοβαρέ αντιρρήσει όσον αφορά τα τυπικά εμπόδια. Αυτά βέβαια μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά πρέπει κυρίω να λύσουμε τα πολιτικά προσκόμματα, τα πολιτικά εμπόδια, του πολιτικού περιορισμού να μην έχουμε υποκειμενικές αξιολογήσεις σε κάτι που επιθυμούν ένα εκατομμύριο πολίτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σέπλιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μίλησαν μέχρι τώρα. Θα ήθελα να καταστήσω κάτι απολύτω σαφέ. Είμαι υπέρ τη πρωτοβουλία των πολιτών. Μπορεί αυτό που θα πω να σα ακουστεί αρνητικό, αλλά είναι ένα είδο τεστ. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται. Καταρχή, δεν σημαίνει ότι όλες οι πρωτοβουλίες θα είναι δημοκρατικές ή ευρωφιλικές. Αν αυτό δημιουργεί συζήτηση, καλώς μερικές πρωτοβουλίες πιθανότητα θα είναι ευκαιρία για λαϊκισμούς. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεύτερο, αν ο στόχος πρωτοβουλίας είναι να επεκτείνει την αίσθηση της ιδιοκτησίας της Ένωσης, οι μη κυβερνικέ οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών δεν νομίζω ότι αυτό θα με οδηγήσει σε μεγαλύτερη ε, ταύτιση ενδέχεται έτσι να πάρουν μέρος περισσότερα άτομα, αν πούμε για την κοινωνία των πολιτών. Αλλά αν αυτό θα περάσει στην ευρύτερη κοινωνία, δεν έχω πιστεί. Δεν έχω πιστεί ακόμη. Τρίτο, χρειαζόμαστε φίλτρα. Για μην έχουμε ενοχλητικές ή επιπόλαιες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να έχουμε επίγνωση ότι αν η γραμμή είναι πολύ χαμηλή, χαμηλά, θα έχει καταστροφικέ συνέπειε. Αν είναι πολύ ψηλή, τότε μπλοκάρεται εντελώ η όλη διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, οι πρώτε πρωτοβουλίε θα είναι πάρα πολύ κρίσιμε προκειμένου να οριστεί το πολιτιστικό πλαίσιο. Και την πιο καλή μέθοδο να παρακολουθούμε, να δημιουργηθεί ένα ιστορικό κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή τις πρώτες πρωτοβουλίες. Και τέλος, μια θεωρητική παρατήρηση. Ουσιαστικά εδώ αναμειγνύομαι αντιπροσωπευτική και άμεση δημοκρατία. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος αυτού. Ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα και αντιρρήσει υπάρχουν για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Πάντως η άμεση δημοκρατία και αυτή δημιουργεί προβλήματα. Να έχουμε επίγνωση του γεγονότος και να μην παρασυρώμαστε από εύκολου ενθουσιασμούς. Επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ του μέτρου, αλλά να έχουμε υπόψη μα ότι μπορεί να υπάρχουν και αρνητικέ πλευρέ. Πρόεδρο. Ο Σνάιφος Μπρόγκς. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία των πολιτών είναι μια πολιτική συζήτηση που κάνουμε και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, σε συνένεση. Όμως, αν από πριν πούμε ότι δεν θέλουμε συνένεση αλλά θέλουμε να συνάδουν πάντα οι πρωτοβουλίες με τις ευρωπαϊκές αξίες, τότε δεν είναι τόσο πολύ μια συζήτηση, είναι μια προκαθορισμένη συζήτηση. Και το είπαμε και σήμερα το πρωί, ότι δεν θέλουμε λαϊκισμό, δεν θέλουμε ε, καταστρεπτικές πρωτοβουλίες. Πρέπει λοιπόν να ελέγχονται οι πρωτοβουλίες αυτές. Επίσης μιλάμε για την ε, άμεση δημοκρατία. Όμως εδώ δεν έχουμε αυτό. Γιατί όταν θα έχουμε το 1 εκατομμύριο υπογραφές, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί παρόλα αυτά να πει μπράβο, ευχαριστούμε πολύ, αλλά εμεί δεν θα προχωρήσουμε με την πρωτοβουλία αυτή. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κάπω αλλιώ πρέπει να λέγεται. Αναφορά θα πρέπει να λέγεται και όχι πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Μέντες δίγω τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω σήμερα, αλλά βλέπετε με τις πτήσεις δεν μπορούμε πάντα να είμαστε στην ώρα μας. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω εδώ δύο παλιούς φίλους που μου φαίνονται βέβαια τόσο νέοι δεν μπορώ να πω ότι είναι παλιοί φίλοι κανενός γιατί μου φαίνονται φοβερά νέοι και ο Μέγερ και η κυρία Κάφμαν. Τους ξέρω από τότε που είχαμε τις συνεδριάσεις μας ε, τις συνέλευσει για το μέλλον της Ευρώπης και θυμάμαι ότι ο Γιώργεν Μέγερ ήταν ένας από αυτούς που ανέλαβε την πρωτοβουλία για το σχέδιο αυτό της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών με τον Λαμασούρ και την ε, Σίλβια βέβαια Κάφμεν η οποία στην προηγούμενη θητεία είχε κάνει έκθεση για αυτό το θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που σας βλέπω εδώ και τους δύο. Πρόεδρε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τώρα που μιλάμε για αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών το εξή. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, και το λέω πάντα στους φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο, είναι μια κοινότητα δικαίου. Άρα δεν μπορούμε να εφεύρουμε διαφορετικές διαδικασίες από αυτές που προβλέπονται ήδη στις συνθήκες. Η αντιπροσωπευτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι εμείς έχουμε εκλεγεί σε εκλογές που λαμβάνουν χώρα κάθε πέντε χρόνια. Οπότε ούτε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ούτε με τίποτα άλλο δεν θα αντικαταστήσουμε την συμμετοχική ε, δημοκρατία ε, με κάτι άλλο. Δεν αντικαθίσταται αυτό με τίποτα. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι ένα θέμα τήρησης των συνθήκων. Οπότε, κοινότητα δικαίου είπαμε. Κατόπιν τούτου φτάνουμε και στο επόμενο, ότι η νομοθετική πρωτοβουλία δεν μπορεί να καταλήξει σε νομοθεσία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκτός δικαίου για να φτάσουμε σε αυτήν την νομοθετική ρύθμιση. Γιατί έτσι λένε οι συνθήκες. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα ε, κατά των αρχών και των αξιών που αναφέρονται στη συνθήκη. Και θα σας το δείξω με ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να συμβεί. Α πούμε ότι έχουμε ένα εκατομμύριο, ή δύο εκατομμύρια υπογραφές που ζητάνε να ξανέχουμε τη θανατική ποινή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο εκατομμύρια, έτσι το ζητάνε. Ωραία, το ζητάνε. Στο άρθρο 2 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και αρέχει νομικά ε, αξία και βάρος, λέει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι βασική αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, όσα εκατομμύρια υπογραφές και αν έχουν συγκεντρωθεί για κάτι τέτοιο, εφόσον δεν πρόκειται για αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να καταδικάσει σε θάνατο, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοια πρωτοβουλία. Και πρέπει να πούμε στους υπογράφοντες, ε, εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να τους πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να νομοθετήσει για κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι πότε τους το λέμε. Τους το λέμε στην αρχή της διαδικασίας ώστε να μην κάνουν τον κόπο, να μην ξοδέψουν χρήματα για να προκαλέσουν κάτι το οποίο δεν θα καταλήξει πουθενά ή τους το λέμε στο τέλος. Περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται περί του ότι κάποιος θα τους υποστηρίξει, δεν θα τους υποστηρίξει. Το θέμα είναι να τους λέμε την αλήθεια, πώς έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό το θέμα δεν έχω καταλήξει. Δεν ξέρω ο έλεγχος πρώτα απ' όλα από ποιον θα γίνεται. Όμως απορρίπτω το αγγλοσαξονικό αυτό επιχείρημα που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ομάδα υπαλλήλων. Δεν συμφωνώ. Ο κύριος Μπαρόσο που ήταν πρωθυπουργό, υπουργό, τι είναι, ο κύριος Αλμούνια που ήταν γενικό γραμματέα ε, στο Σελιστικό Κόμμα, υπουργέ κτλ. Όλοι αυτοί είναι πολιτικοί, δεν είναι υπάλληλοι. Ναι, σα το λέω και εσά, δεν είναι υπάλληλοι. Είναι πολιτικοί που εμεί εκλέξαμε. Και άρα εμεί μπορούμε και πρόταση μορφή. Και θυμηθείτε τι έγινε με την Επιτροπή του Σαντέρ. Άμα θέλουμε, κάνουμε μια πρόταση μορφή και πάνε. Δεν είναι δυνατόν Κάποιοι υπάλληλοι λένε ορισμένοι να παίρνουν μια τέτοια απόφαση. Ναι, αλλά εμείς και οι συνθήκες τους δίνουν το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας. Οπότε έχει νόημα να είναι η Επιτροπή εκείνη η οποία τελικά να ετοιμάσει μια νομοθετική πρόθεση που να βασίζεται στο αίτημα των πολιτών με την πρωτοβουλία τους. Μου φαίνεται λογικό αυτό. Τώρα όπως είπα και πριν, Μπορεί να υπάρχει και άλλη μέθοδος, πιο ενδιαφέρουσα, πιο δημοκρατική ή πιο κατάλληλη. Αλλά επιμένω στο αρχικό μου επιχείρημα, Πρόεδρε. Στον κόσμο πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να τους δημιουργούμε φοβερές προσδοκίες και να τους πούμε «Α, θα υπάρξει άμεση δημοκρατία». Όχι, είναι ένα μέσο αποτελεσματικό, συγκεκριμένο η πρωτοβουλία αυτή που θα επιτρέψει στον κόσμο να συγκεντρώνεται και να, βασίζει, να στηρίζει από κοινού μία ιδέα. Οι Ευρωπαίοι έχουν μάθει να συγκεντρώνονται γύρω από ιδέε, γύρω από προγράμματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και με αυτό θα τελειώσω, ότι η θεσμική μέθοδος των συνθήκων, όλες οι βασικές αρχές της κοινότητας δικαίου, μπαίνει στην πάντα επειδή έχουμε τώρα μια νέα πρωτοβουλία και εφαρμόζονται άλλες αρχές αυτή. Όχι. Πρόεδρε, το χειρότερο Εντάξει, θέλουμε φυσικά να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες. Μας έχει γίνει έμονη ιδέα. Αλλά το χειρότερο δεν είναι να τους φοβόμαστε. Το χειρότερο είναι να μην τους λέμε την αλήθεια, να μην τους λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο σε προσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου, θέλω και εγώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Στην Ιταλία έχω μια καλή εμπειρία και από διάφορα ε, δημοψηφίσματα με αρνητικό χαρακτήρα και πρωτοβουλίε πολιτών. Όσον αυτό το έλεγχο του παραδεκτού ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντομα. Όσο πιο σύντομα, στην αρχή. Στην αρχή. Πριν καν ε, συλλεγούν, συγκεντρωθούν υπογραφές, θα έλεγα. με στο χρονοδιάγραμμα που είπε ο συνάδελφος Μέντες Δεβίγκο. Μπορεί κάποιο να πει α, να φύγει η Γαλλία από την Ένωση, παραδείγματο χάρη. Ε, ε, ε, δεν μπορεί ε, οποιοδήποτε έτοιμο... ένα έτοιμο όπως αυτό να γίνει αποδεκτό. Ο αριθμός τώρα αυτών που προτείνουν μια πρωτοβουλία. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία που τελικά θα πρέπει να πιάσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες από ενορισμένο αριθμό χωρών. Αρκετές χώρες. Τώρα θα είναι 7 χώρες ή 5 ή παραπάνω, δεν ξέρω. Αρκετές χώρες. Μία πρωτοβουλία σημαίνει επαφές μεταξύ των χωρών. Μία πρωτοβουλία που δεν μπορεί από την αρχή να συγκεντρώσει 7 άτομα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αρχικό νούμερο, αν δεν καταφέρει τουλάχιστον έχει τουλάχιστον 10 πολίτες από διαφορετικές χώρες μέλη, αυτό σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. Ένα άλλο θέμα σοβαρό είναι η ταυτοποίηση. Για να είναι σοβαρή μια πρωτοβουλία πρέπει να είναι σοβαρή. Άρα δεν πρέπει να έχουμε δύο φορές να υπογράφει το ίδιο άτομο. Να μην υπάρχουν ψευδείς υπογραφές που είναι εύκολο να γίνει αυτό αν δεν υπάρξει έλεγχος. Να γίνει έλεγχος ότι ο τάδε πολίτης επειδή η πρωτοβουλία είναι σοβαρή ζητάει αυτό. Γιατί να μιλάμε γενικά για όλες τις χώρες αυτό θα δυσκολέψει τα πράγματα. Έχουμε εμπειρίε στις χώρες μας. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε κάθε χώρα να ελέγχει τη σοβαρότητα και το πόσο ε, γνήσεις είναι οι υπογραφές. Αν δεν φτάσουν το 1 εκατομμύριο υπογραφές, τι γίνεται. Πού είναι το πρόβλημα θα μπορούσε το κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια των διακριτικών εξουσιών του θα μπορούσε να το κάνει. Υπάρχει ένα δικαίωμα αναφοράς από εκ μέρους ενός ατόμου. Άρα κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσε ένα τέτοιο αίτημα που δεν φτάνει το 1 εκατομμύριο να μπορεί να μετατραπεί σε ένα είδος αναφορά. ηλικία. Μόνο η Αυστρία προβλέπει 16 έτη ηλικία. Αν ήταν ποδόσφαιρο θα λέγαμε 26-1. Κατά τη γνώμη μου το 16 είναι δύσκολο να το δεχτούμε. Μία ερώτηση τώρα. Υποδείξεις είναι όλα αυτά και ερώτηση προς τους εμπειρογνώμονες αν το αντικείμενο της πρωτοβολίας θα μπορούσε να είναι μια τροποποίηση των συνθήκων ή όχι. Προσωπικά θα έλεγα γιατί όχι. Αλλά έχουμε το άρθρο 225. Πώς μπορούμε να το υπερπηδήσουμε. Ναι, το κοινοβούλιο έχει τις εξουσίες και οι πολίτες έχουν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο ένα είδος ρόλου τόνωσης ως προς την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία με βάση ένα συγκεκριμένο άρθρο να κινήσει μια διαδικασία τροποποίησης των συνθηκών. Αυτό όμως δεν προβλέπεται για τους πολίτες, άρα υπάρχει κάποιο όριο νομικό που είναι δύσκολο να υπερπηδηθεί κατά τη γνώμη μου. Το θέτω ως ερώτηση προς τους εμπειρογνώμονες. Μιλάω κι εγώ τώρα ως μέλος, δεν μιλάω ως πρόεδρος, ως μέλος μίλησα της Επιτροπής. Και τώρα παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο κύριος Τενραϊρά. Um, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση που παρακολούθησα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή για να κάνω κάποια σχόλια σε τρία σημεία. η ιδέα της Επιτροπής των Πολιτών, το παραδεχτό και η επαλήθευση των υπογραφών. Για το πρώτο, η Επιτροπή αυτή των πολιτών δεν είναι ιδέα της Επιτροπής, κυκλοφορεί γενικά στο Κοινοβούλιο. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Διότι θα μπορούσε να βοηθήσει να προχωρήσει καλύτερα η διαδικασία, να υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση και να πρόκειται για μια σοβαρή πρωτοβουλία που έχουν σκεφτεί οι πολίτες καλά. Και έτσι θα ελαφρύναμε κάπως τους άλλους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνουν μετά. Οπότε είμαστε ευέλικτοι και την εξετάζουμε με ενδιαφέρον την ιδέα αυτή. Αυτό φυσικά που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και λοιπά από τους πολίτες και όλοι αυτοί πρέπει να ξέρουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν την Επιτροπή των Πολιτών. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν. Για το θέμα του παραδεκτού των πρωτοβουλειών. Θέλω και εδώ να τονίσω ποιο είναι το κείμενο της Επιτροπής και τι υπάρχει στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Δεν είναι προσπάθεια να υπάρξει μια κύρωση. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο αυτό. Όταν ε, μιλάμε για τους ελέγχους που θα γίνονται, δεν θα γίνονται υποκειμενικά. Ο έλεγχος σημαίνει αυτό που λέει και η λέξη, έλεγχος. Αλλά όχι με στόχο να κάνουμε λογοκρισία. Σε μια ακρόαση Ε, είχα δώσει ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι οι πολίτες ζητάνε στι Ολομέλειες να πηγαίνουν οι ευρωβουλευτές ντυμένοι μπλε με κίτρινα στεράκια. Ε, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να είναι σοβαρέ οι πρωτοβουλίες που γίνονται. Και θέλω να πω στον κύριο Μέντες Δεδίγο η πρωτοβουλία αυτή που έφερε σαν παράδειγμα για τη θανατική ποινή. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να καταγραφεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εμείς δεν θα δώσουμε συνέχεια σε μία πρωτοβουλία η οποία αντιτίθεται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα συζητήσουμε καν το αν υπάρχει νομική βάση για να προταθεί ένα τέτοιο μέτρο. Από την αρχή πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν θα καταγραφεί και δεν θα μπει στην ιστοσελίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον αντιτίθεται στι ευρωπαϊκέ αξίε. Δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο είναι λογοκρισία. Είναι μια πολιτική εκτίμηση. Τώρα συμμετέχουμε στις συζητήσεις που γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και ακούμε όλες τις ιδέες όσον αφορά τον ε, έλεγχο των υπογραφών. Όλες τις ιδέες λοιπόν τις καταγράφουμε, τις προσέχουμε. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες σας και σε ένα βαθμό κάπως αυτό αντικατοπτρίζεται στο κείμενο του Συμβουλίου, το οποίο στα κριτήρια προσθέτει και ένα άλλο που είναι ότι δεν πρέπει να καταγράφεται μια πρωτοβουλία εφόσον είναι εκτός πλαισίου συνθήκων. Άρα λοιπόν είναι ένα βήμα μπροστά παραπάνω. Αλλά δεν είναι μια πραγματική δοκιμή για την νομική βάση. Μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την ιδέα και να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε ένα κριτήριο βάσει του οποίου να μπορούμε ξεκάθαρα να αποφασίζουμε ότι είναι εκτός πλαισίου συνθήκων μια πρωτοβουλία. Και έτσι θα απλοποιηθεί κάπως η διαδικασία. Παράδειγμα, ασφαλιστούμε ότι έρχονται πρωτοβουλίες για να αλλάξει η κατανομή των Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εκτός πλαισίου συνθήκων, είναι εντός πλαισίου συνθήκων. Οπότε θα έπρεπε να καταγραφεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Και μετά θα πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει νομική βάση για να κάνει νομοθετική πρόταση για αυτό το θέμα. Αν αλλάξουμε όμως το κείμενό μας, μπορούμε να βρούμε τρόπο από την αρχή να λέμε στους πολίτες ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζει η Επιτροπή και ότι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την πρωτοβουλία να αποφασίζει για την κατανομή των Ευρωβουλευτών στο σώμα. Οπότε από την αρχή να απορριφθεί αυτή η πρωτοβουλία. Πάντως είναι σημαντικό να υπάρχει από την αρχή μια πλήρης νομική εκτίμηση. Και επιμένω σε αυτό. Τέλος, για τους ελέγχους. Αυτή είναι μια συζήτηση που βέβαια κυρίω γίνεται ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα ελέγχου. Πάντω θέλω να κάνω κάποια σχόλια και εγώ για να διευκρινίσω λίγο αυτό το σημείο. Πρώτον, οι έλεγχοι γίνονται τυχαία, δειγματοληπτικά. Δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος. Κανένα δεν περιμένει τα κράτη-μέλη να καθίσουν και να ελέγξουν όλες τις ε, υπογραφές. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν τις υπογραφές αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε, λέμε έλεγχος υπογραφών, αλλά δεν είναι αυτό που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε online συλλογή υπογραφών, δεν θα είναι πραγματικά υπογραφές, θα είναι μια επιβεβαίωση. Κάποιος με το email του θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία. Δεν ελέγχουμε λοιπόν πραγματικά τις υπογραφές, ελέγχουμε τα στοιχεία του ατόμου. Αν τα στοιχεία του ατόμου κολλάνε, δηλαδή όντω υπάρχει ένα άτομο με αυτό το όνομα που ζει σε αυτή την πόλη και γεννήθηκε τότε κτλ τότε εντάξει. Θεωρούμε ότι πράγματι αυτός έχει βάλει την υπογραφή του. Τέτοιου είδου ελέγχου κάνουμε. Το πρόβλημα είναι βέβαια βάσει τίνος πράγματος ελέγχουμε. Τα κράτη-μέλη μα έχουν πει μέχρι τώρα ότι ο μόνος τρόπος που έχουν για να ελέγξουν είναι να πάνε σε βάσει δεδομένων που συνδέονται με έγγραφα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουν πού να ψάξουν. Άρα πρέπει να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται και που τεχνικά μιλώντας είναι δύσκολη. Εμείς ευχαρίστως να βοηθήσουμε, αλλά ήθελα να σας διευκρινίσω πώς έχει η κατάσταση. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και ο εκπρόσωπος Συμβουλίου, ο κύριος Um, ευχαριστώ. Ορισμένα τα είπε και ο κ. Σαστέλ της Βελικής Προεδρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα, ευχαριστώ. Εισηγητές και εμπειρογνώμονες για την εντελεχή εξέταση του θέματος. Όπως είπε ο υφυπουργός μου, η Βελική Προεδρία μοιράζεται την φιλόδοξη στάση του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν με, την, με τον στόχο να φτάσει σε πρώτη ανάγνωση πριν από το τέλος του έτους. Επίσης θεωρεί ότι η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να είναι εγγύς των πολιτών κάτι που είναι σαφές και από την θέση του Συμβουλίου. Στην κοινή θέση της 14ης έκτου. Επίσης, είναι σημαντικό οι πρωτοβουλίες αυτές να είναι αποτελεσματικές και υλοποιήσιμες. Υπάρχουν και ορισμένα τεχνικά θέματα, όπως ελέγχθη προηγουμένω, στα οποία θα εγκύψουν οι χώρε μέλη, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία δίνουν οι πολίτες. Η συνεργασία υπήρξε εξαιρετική με τους τέσσερις εισηγητάς και αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχιση του διαλόγου έτσι ώστε να φτάσουμε σε πρώτη ανάγνωση όπως είπα πριν από το τέλος του έτους. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο για να απαντήσουν οι δύο προσκεκλημένοι μας και η συγγήτρια κυρία Γκουρμάη έχουν ζητήσει το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Σας προεδοποιώ στο μεταξύ ήρθε και ο Μαρτίνες και δεν θέλουμε να το κάνουμε περιμένει για να περάσουμε και στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ λοιπόν να είστε λακωνικοί. Ο Σάνφος Μέρσα Σμιτ, πρώτος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Δεν πήρα απάντηση στην ερώτησή μου. Έχουμε ένα σωρό κανονισμούς στη συνθήκη που περιορίζουν την Κομισιόν από το να υποβάλει πρωτοβουλίες. Γιατί στη συγκεκριμένη πρόταση αυτή της Κομισιόν έχουμε αναφορά όχι μόνο σε άρθρα, αλλά σε συγκεκριμένα κριτήρια, μόνο στις αξίες δηλαδή. Και δεν μιλάω για τη θανατική ποινή, περισσότερο θα είναι κατά, τουλάχιστον στο Ευρωκοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη, α πούμε, κάποιο ε, θέτει να αμφιβόλο την αρχή της αναλογικότητα ή της επικουρικότητας Αυτό θα είναι παραδεκτό μεν, αλλά μη εφαρμόσιμο στην πράξη. Δεν μπορεί να το προτείνει αυτό η Κομισιόν. Γιατί έχουμε λοιπόν περιορισμούς που αποκλείουν προτάσεις που στηρίζονται στις αξίες και όχι όλα τα άλλα κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου να δράσει η Ένωση. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μου. Και γιατί δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα άρθρα, όταν μιλάμε για αξίες είναι το άρθρο 6 που αναφέρεται στη χάρτα που ανάφερε ο κύριος Δεβίντε, είναι το άρθρο 2 που αναφέρεται στις αξίες. Για τι πράγμα μιλάμε. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, για το τμήμα 3. Με ποια βάση θα αξιολογήσουμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Ντάφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που έλειψα από τις συζητήσεις μέχρι τώρα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ και η κυρία Κάφμαν και ο κύριος Μέγερ που είναι εξέχοντα τέος ε, μέλη εδώ. Έχουν ε, δώσει μάχες στο παρελθόν μαζί. Τις δώσαμε. Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να μείνει εκτός της διαδικασίας ε, ελέγχου του παραδεκτού των πρωτοβουλειών. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ή να τη βάλουμε εμεί στη θέση όπου είναι και κριτής και κρινόμενος, που κρίνει δηλαδή το παραδεκτό και συγχρόνως αποφασίζει για το τέλος της διαδικασίας. Τι θα κάνει δηλαδή με την πρωτοβουλία, την κάθε πρωτοβουλία. Αν πολιτικά δηλαδή θα προχωρήσει η πρόταση ή όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο περίπλοκο να πούμε κατά πόσο μια πρωτοβουλία παραβιάζεται τη συνθήκη όχι. Αν εμένα με ρωτήσουν, μέσα σε ένα τέταρτο έχω έτοιμη την απάντηση αν είχα τον υπολογιστή μου, θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αμέσω. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας επιστήμονας. Χρειάζεται απλώς να γνωρίζει κανείς καλά το εύρος των αρμοδιοτήτων και τα περιολοκλήρωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κάνουμε μια περίπλοκη διαδικασία τώρα όταν μιλάμε για επιτροπές σοφών, που στο κάτω-κάτω θα είναι και ακριβή μια τέτοια επιτροπή σοφών. Θα πρέπει να πληρώνεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ή όταν λέμε η επιτροπή να είναι εκείνη η οποία θα αποφασίζει για το ξεκίνημα της διαδικασίας ή όχι. Είναι λάθος αυτό. πρέπει να αποφασίσουμε επί της αρχής. Θέλουμε κάτι τέτοιο ή όχι. Ο κύριος Κασίνη περιγράφει πολύ ρεαλιστικά την Ιταλική εμπειρία. Σωστά. Όντως θα υπάρχουν πολλές ψεύτικες υπογραφές ή διπλές υπογραφές. Το τέλος δεν ξέρω αν πειράζει αυτό τόσο πολύ. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ψεύτικων υπογραφών, τουλάχιστον να μην είναι πολλές. Πάντως, αν υπάρχει ένα νούμερο που είναι γύρω στο ένα εκατομμύριο υπογραφών και οι οποίοι θέλουν νομοθετική πρωτοβουλία, Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να το λάβουν υπόψη τους. Μην είμαστε πολύ γραφειοκράτες, να είμαστε ρεαλιστές και να επιτρέψουμε την συνέχιση της διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό. Αν υπάρχει μια πρωτοβουλία που θέλει περισσότερες δαπάνες, η μείωση δαπανών, αυτό παραβιάζει την πολιετή δημοσιονομική συμφωνία. Τι λέμε τότε. Στο email που έρχεται από μια ομάδα πολιτών οι οποίοι θέλουν να αλλάξει εκεί κάτι. Εδώ θα ήθελα να με βοηθήσετε συγητέ ή όσοι τέλος πάντων έχουν εμπειρία πάνω σε τέτοια θέματα να μου πείτε τι κάνουμε τότε. Ίσως θα μπορούσαν να αποκλείονται τέτοιες πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα. Θέλω όμως την άποψή σας. Τέλος. Όπως γνωρίζετε, στην πρότασή μου για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας Μιλάω για μια εκλογική αρχή η οποία θα εποπτεύει την πανευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε περιθώριο για μια τέτοια ανεξάρτητη εκλογική αρχή η οποία να επαληθεύει την αξιοπιστία μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Εάν ναι, αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε την ε, παρεμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Απαντήσεις δυστυχώς ο χρόνος είναι ελάχιστος πια. Παρακαλώ τους δυο προσκεκλημένους μας, τον κύριο Μάγερ και την καθηγήτρια κυρία Κάουφμαν. Oh, ευχαριστώ πρώτα για τις ε, πολλές και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Άκουσα ότι η πρώτη ανάγνωση του κανονισμού θα προβλέπεται προ του τέλους του έτους. Δηλαδή 7,5 χρόνια. Ωστόσο, από τότε που ε, πέρασε η πρόταση αυτή στη συνταγματική συνέλευση. Αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας κύριε Κατσίνη ότι η εξέταση του παραδεκτού θα πρέπει να γίνεται στην αρχή. Και γι' αυτό έκανα την πρόταση μετά από 5 ή το πολύ 10.000 υπογραφές να γίνεται μια εξέταση και μετά να καταχωρίζεται η πρωτοβουλία. Ο φίλος μου η Νίκο Μέντες ήδη στο Προεδρείο της Συνταγματικής Συνέλευσης ως μειοψηφία τότε ο ίδιος είχε υποστηρίξει την πρωτοβουλία και έχει δίκιο που λέει ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν υποκαθίσταται αλλά εμπλουτίζεται με ένα σημαντικό στοιχείο άμεσης δημοκρατίας. Και σε ό,τι αφορά τις αξίες έφερε στο παράδειγμα της θανατικής ποινή. Όλα όμως περιλαμβάνονται στο έγγραφο που ήδη τότε στην πρώτη συνέλευση είχαμε επεξεργαστεί μαζί στον χάρη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ δεν θα, δια... δεν θα μαλώσω τώρα εδώ αν θα πρέπει να είναι το άρθρο 2 ή το 6 αλλά είναι ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το έγγραφο που διαλαμβάνει τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντριου Νταφ, που επιθυμεί να βγάλει απ' έξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εξέταση του παραδεκτού. Μου φαίνεται αξιοσημείωτη αυτή η πρόταση, διότι αλλιώ η ε, ε, Κομισιόν μπαίνει σε ένα δίλημα. Αφενός δηλαδή να εξετάζει το παραδεκτό, αφετέρου να είναι υποχρεωμένη να εκρίνει εάν θα δώσει συνέχεια σε μια πρωτοβουλία ή όχι. Για τον λόγο αυτό, εγώ έχω κατανόηση και δέχομαι αυτό το Συμβούλιο των Σοφών με την προστίκη όμως ότι εφόσον αυτοί που ναι στο παραδεκτό, η απόφαση τους αυτή θα πρέπει να είναι τελεσίδικη. Εάν πουν όχι, θα πρέπει να επανεξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διότι με τον τρόπο αυτό ανοίγεται πλέον η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν όμως πούν ναι οι σοφοί, τότε αυτό θα πρέπει να είναι τελεσίδικο. Και τότε θα πρέπει εκεί να λύγει η εξέταση του παραδεκτού. Ο κύριος Χέφνερ έκανε μερικέ ερωτήσει. Θα απαντήσω σε τρει από αυτέ ή τέσσερι. διαφάνεια σχετικά με τους υποστηρικτές και χρηματοδότηση. Αυτή η διαφάνεια θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη στην καταχώρηση. Τότε αρχίζει λοιπόν η προσπάθεια, αρχίζουν οι συλλογές των υπογραφών και εκεί θα πρέπει να είναι σαφές πλέον ποιο ενδεχομένως υποστηρίζει και χρηματοδοτικά την πρωτοβουλία. Επίσης ο συναδελφός μου τόνισε ότι στην επαλήθευση και εξέταση των επιμέρους υπογραφών δεν θα πρέπει να ισχύουν οι δυνατόν διαφορετικές ρυθμίσει στις χώρες μέλη. Αυτό μου φαίνεται επιθυμητό ως στόχος. Αλλά για την περίπτωση που αυτό δεν γίνει δεχτό από το Συμβούλιο, θεώρησα εγώ ότι τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βγει και να πει καθαρά τι θέλει. Να πει για παράδειγμα ότι αυτή η ανοησία περί της ε, ανακοίνωσης του της καταγραφής δηλαδή του αριθμού της προσωπικής ταυτότητας ή του προσωπικού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης, ότι αυτά είναι ανοησίες και να, παρα... και να μείνουν εκτός. Τώρα, η μνήα της νομικής βάσης που διαλαμβάνεται στο έγγραφο ε, των εισηγητών. Μου φαίνεται και αυτό ότι είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολική επιβάρυνση δηλαδή για εκείνους οι οποίοι θα ε, προχωρήσουν σε μια πρωτοβουλία γιατί θα χρειαστεί αμέσως να αναζητήσουν νομικές συμβουλές. Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει από το Συμβούλιο των Σοφών. Γιατί οι, οι ίδιοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να πούν ακριβώς ποια είναι η νομική βάση. Το ερώτημα τώρα που τέθηκε από πολλούς ότι δηλαδή αντικείμενο της πρωτοβουλίας θα μπορεί να είναι και η περαιτέρω εξέλιξη των συνθήκων. Η κυρία Γέτα Μάκη το υποστήριξε, αλλά εξέφρασε κάποιε επιφυλάξει ο πρόεδρο, τι οποίε σχολιάζω. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγωγός 4 τη συνθήκη, η πρωτοβουλία εξυπηρετεί την εφαρμογή των συνθήκων. Το ίδιο, και εγώ τήρησα ακριβώ την διατύπωση αυτή, το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 225 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο το ίδιο έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει η πρωτοβουλία για την τροποποίηση των συνθήκων. Τα λέει αυτά το άρθρο 48. Όμως, εάν το Κοινοβούλιο επιλέξει την οδό του άρθρου 225, δεν πράττει αυτό, αλλά κάνει ακριβώς ό,τι και μια πρωτοβουλία πολιτών, δηλαδή υποβάλλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει τέτοια πρωτοβουλία νομοθετική ρυθμιση. Πρόκειται λοιπόν για εξίσωση του άρθρου 11 πρωτοβουλία πολιτών και 225 συνθήκης υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ εδώ θεωρώ ότι τίθεται το θεμελιώδες ερώτημα. Δεν σημαίνει πραγματική ζωντανή δημοκρατία να εξελίσσεται κιόλα και σε ό,τι αφορά τη θεσμική της βάση. Πρέπει όμως να λεχθεί στους πολίτες εφόσον θέλετε να ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε το άρθρο 48 που προβλέπει κύρωση και από τις 27 χώρες μέλη. Και τότε ορισμένοι πολίτες τουλάχιστον θα αντιληφθούν ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που ασφαλώς δεν πρόκειται να κυρωθούν από όλες τις χώρες μέλη. Το γνωστό παράδειγμα της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει η Γαλλία. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίσει και να το πει στους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να αποφασίσουν διαφορετικά. Μία διατύπωση ωστόσο που προέκυψε από διάφορες συζητήσεις και με το Συμβούλιο είναι ότι το θέμα της πρωτοβουλίας δεν θα πρέπει να κείται εκτός συνθήκων. Η τροποποίηση όμως των συνθήκων σύμφωνα με το άθρο 48 είναι μέσα στις συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν οι συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ήδη εδώ μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει ως βάση για να το δεχτεί. Επιμένω όμως ότι η πρόταση της Σίλβια Ιβόν Κάουφμαν μια νέα διαδικασία ενδεχομένως μέσω του ε, κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες με μια τέτοια πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι καλή ε, η ιδέα αυτή, αλλά δεν είναι εναλλακτική επιλογή. Θα πρέπει η πρωτοβουλία να ε, έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στην Κομισιόν και ενδεχομένω σωρευτικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι διαζευτικά. Αυτό θα σήμαινε εμπλουτισμό και όχι απλώ μια κάπως στενόκαρδη υποκατάσταση. Τέλος, στις συνθήκες περιλαμβάνονται πολύ, πολλά συγκεκριμένα πολιτικά ε, πράγματα από την παλιά συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που έχουν διαλυθεί τώρα και στις συνθήκες της Ένωσης που είναι πολύ εύκολο να απορριφθούν διάφορες ε, πρωτοβουλίες πολιτών επειδή δεν είναι απόλυτα σύμφωνες με διάφορες προβλέψεις. Αυτό όμως καλύτερα να μην το κάνετε να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα απέναντι στους πολίτες, να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου και διαμεθοριακά και εν τέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί και να ανδρωθεί ή να γυναικωθεί αν θέλετε και να σηκωθεί και να πει κοιτάξτε δεν το θέλουμε αυτό την απόφαση θα τη λάβουν τελικά οι Κομισιόν, οι εμείς τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα να μπαίνουν τώρα απαγορευτικά γραφειοκρατικά κολλήματα εκ μιας αρχής, αυτό δεν είναι σωστό. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση της Επιτροπής Πολιτών στην αρχή, ας το ξανασκεφτούμε, ας μην είναι προϋπόθεση, ας γίνει μια σύσταση να ιδρυθεί μια Επιτροπή Πολιτών, ώστε να υπάρχει ένα συνομιλητής που θα απαρτίζεται από ε, ανθρώπους που θα προέρχονται από διάφορες χώρες. Εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτό, τότε θα σημάνει βέβαια το τέλος της πρωτοβουλίας, έστω. Αλλά είναι και πολύ πιο φιλική η συνδιαλλαγή με τον τρόπο αυτό με τους πολίτες. Κάουφμαν. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση και βεβαίω εξακολουθούν να ακούονται διάφορες απόψεις για διάφορα θέματα και από παλαιούς συναδέλφους μου, για παράδειγμα Άντριου Ντάφ Η πρωτοβουλία απευθύνεται στην Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει το μονοπόλιο της ανάλυσης πρωτοβουλίας για νομοθετικές ρυθμίσεις. Η αρχή αυτή δεν τροποποιείται. Και η Κομισιόν λαμβάνει, για παράδειγμα, προτάσεις από το Κοινοβούλιο για να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, θα πρέπει τότε να εξετάσει αυτή ποια είναι η νομική βάση. Εγώ θεωρώ ότι η Κομισιόν δεν επιτρέπεται να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή. Αυτό που είναι σαφές εξάλλου είναι ότι σε ό,τι αφορά την εξέταση παραδεκτού θα πρέπει αυτή να είναι μοναχά νομική και διόλου πολιτικού χαρακτήρα. Αυτή η νομική εξέταση του παραδεκτού θα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη βάση. Εδώ νομίζω ότι η συμπλήρωση που κάνει το Συμβούλιο στην πρόταση της Κομισιόν στις, του, στις γενικές του κατευθύνσεις είναι σωστή. Ότι δηλαδή θα πρέπει να εντάσσεται την πρωτοβουλία αυτή, το θέμα της δηλαδή, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και να αναφέρεται στις αξίες του άρθρου 2. Εφόσον τηρηθεί αυτό, για μένα είναι σαφές ότι μένει πια μόνο η νομική αυτή εξέταση. Και οι διάφορε ανησυχίε, για παράδειγμα και του κ. Σέφλιν, ότι ενδέχεται να γίνει κατάχρηση τη πρωτοβουλία των πολιτών, με τον τρόπο αυτό έρεται το ενδεχόμενο αυτό. Το παράδειγμα του Μέντε Στεβίγκο με τη θανατική ποινή είναι εξαιρετικό. Διότι από την αρχή είναι προφανέ ότι η Κομισιόν δεν χρειάζεται να ασχοληθεί. Ε, χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα λέει αυτά. Επιστρέφεται στην αποστολέα η ε, πρωτοβουλία. Επίσης έγιναν, τέχθηκαν διάφορες ερωτήσεις από τον Γκέραντ Χέφνερ. Θα αναφερθώ εγώ σύντομα σε αυτό. Το ερώτημα ήταν πώς μπορεί να εμποδιστεί να μπουν πλήρωνε υπογραφές σε μια πρωτοβουλία. Εδώ η πρόταση μου φαίνεται σωστή, στο παράρτημα 3 δηλαδή, δηλαδή στο άρθρο 7 λέει σαφώς ότι δηλώνει ο υπογράφων ότι έχει υπογράψει, υπογράψει μόνον άπαξ. Αυτό είναι μια βάση εμπιστοσύνη από την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτά στο έγγραφο τη ε, συμμετοχή. Σε ό,τι αφορά την διαφάνεια για τη χρηματοδότηση, η πρόταση Κομισιόν είναι σωστή. Βέβαια, μπορεί να σκεφτεί κανένας και να διαρωτηθεί αν είναι και επαρκές να, γίνει, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης από την αρχή. Είναι δυνατόν, διό, είναι δυνατόν στην πορεία της συλλογής υπογραφών που ας πούμε ότι θα διαρκέσει 18 μήνες κάποιοι να ε, βάλουν χρήματα σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ίσως όχι στην αρχή, αλλά α πούμε μετά από έξι μήνε. μπορεί μια επιχείρηση ή κάποιος άλλος να αποφασίσει να βάλει ε, κάποια λεφτά. Άρα η καποιο αλλο να είναι δεδομένη σε όλη τη διάρκεια της συλλογής υπογραφών. Και όχι μόνο στην αρχή. Τώρα, τα στοιχεία των υπογραφώντων. Σαφές. Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκότητα, υπογραφή. Αυτά αρκούν. Τον αριθμό αστυνομική ταυτότητας, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Δεν θα βρείτε κανέναν που να έχει ακριβώς το ίδιο όνομα, την ίδια ημερομηνία γεννήσεως, την ίδια κατοικία. Αυτά δεν γίνονται και θα πρέπει βεβαίως να επιτρέπεται μόνο δειγματοληπτικό έλεγχος και μόνο από τι φορέ μέλη. Δεν μπορεί να γίνει από την Κομισιόν κάτι τέτοιο. Τελευταία παρατήρηση προς την κατεύθυνση του κυρίου Μπράουν που είπε προηγουμένω ότι η πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι άμεση συμμετοχική δημοκρατία, δεν είναι παρά μόνο μια αναφορά με διαφορετικό όνομα. Όχι. Ακριβώς όχι. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών και αυτό που επιδιώκουμε με την πρωτοβουλία πολιτών είναι οι πολίτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα προτροπής όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτροπής σε ανάληψη <clears throat> νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή στο συγκεκριμένο αυτό οι πολίτες έρονται στο ίδιο ύψος με τα θεσμικά όργανα. Είναι κάτι διαφορετικό από το δικαίωμα αναφοράς που γνωρίζουμε από τις συνθήκες. Τα αυτά και μένω, κύριε Πρόεδρε, εν συντομία, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ε, καλή επιτυχία στην υπόλοιπη προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνουμε την πρώτη αυτή φάση με την παρέμβαση της ε, Αντιπρόεδρου κυρίας Γκουρμάη, η οποία σίγουρα θέλει να πει κάτι. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Γκουρμάη. Σύντομα όμως παρακαλώ. Αγαπητοί συναδελφοί, Πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ μεγάλη σημασία. Με την ακρόαση αυτή και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας ιδιαίτερα Σνάιφο Κάουφμαν και επειδή είμαι πρακτική γυναίκα ε, βρήκα πολύ θετικά τα 8 σαφή σημεία που επισημάνατε. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιούργεν. Σας συγχαίρω για το ότι πήρατε σοβαρά το θέμα αυτό. Είχαμε τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια την περασμένη εβδομάδα. Θα γίνει και άλλη συζήτηση. Τώρα αυτό που θέλουμε είναι να γίνει μια καλή έκθεση. Είμαστε μια ομάδα τεσσάρων που δουλεύουμε για το θέμα αυτό. Είμαστε και σε μια διαδικασία εκμάθησης κατά κάποιο τρόπο. Και όπως είπε σωστά ο συνάδελφος από την Ουγγαρία, δεν ξέρουμε τελικά πού θα καταλήξουμε. Είναι μια περιοχή αχατογράφητη εδώ που κινούμαστε. Να πηδήξουμε στο νερό, δεν ξέρουμε τι βάθος έχει το νερό. Ένα σωρό ερωτήματα παραμένουν ακόμα αναπάντητα. Πολλές ωραίες ιδέες ακούστηκαν. Θα τις επεξεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντική επίσης η παρουσία της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από την αρχή. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές πιθανότητες μετά τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας τον Νοέμβριο και ψηφοφορία στο τέλος Νοεμβρίου να έχουμε μια πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια και ένα καλό αποτέλεσμα. Και οι τρεις εταίροι, από ό,τι φαίνεται, δείχνουν ευελιξία, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το, αυτή την αναγκαία συνένεση. Και ας μην ξεχνάμε, για να λειτουργεί η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών, είναι ένα παλιό χρέος που έχουμε έναντι των πολιτών μας. Πέρασε σχεδόν ένα χρόνο από τότε υπάρχει στην ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνας. Και σωστά θα μα ρωτήσουν γιατί να μην χρησιμοποιούμε αυτό το δημοκρατικό εργαλείο, γιατί όχι. Έχουμε λοιπόν σοβαρή ευθύνη. Χαίρομαι που ο Ισπανός συνάδελφος κάθεται δίπλα μου και είναι και άλλοι Ισπανοί συνάδελφοι στην αίθουσα. Οι τρει προεδρίες και η Βελγική και η Ισπανική φρόντισαν να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Είχαμε ότι έγγραφο εργασία στην Ισπανική Προεδρία και δεν ήταν τυχαίο αυτό. Και έγινε και συζήτηση στην Επιτροπή μας. Ποιος θα πάρει την έκθεση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεργάζεται μαζί μας και η Επιτροπή Αναφορών προκειμένου να πετύχουμε, όπως είπα και πριν, μια ισχυρή συνένεση. Την έκθεση θα φροντίσουμε να την έχει τόσο πιο σύντομα γίνεται, με στόχο την πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, η συμφωνία, η τελική, θα πρέπει να στηρίζεται σε ευρία ομοφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο των πολιτικών ομάδων, και μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και οι τέσσερι στην ομάδα μας έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Θα εισακούσουμε και νέες προτάσεις και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Σας διαβεβαιώνω, δεν θα επιβραδύνουμε το βήμα μας. Για να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι υπάρχουμε λόγω αυτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ όλους τους προσκεκριμένους για την παρουσία σας και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, γιατί έχει εδώ κάμποση ώρα ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνας και του ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση, γιατί είχαμε πει να αρχίσουμε στις 11. Το σημείο λοιπόν 11 αφορά την εξελίξη στην Κοζάκ. Συνήθω οι υπεύθυνοι του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην Κοζάκ μετά τη συνεδρίαση της Κοζάκ έρχονται και κάνουν αναφορά στην Επιτροπή. και παρουσιάζουν τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη ΚΟΖΑΚ. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε στη Μαδρίτη, η επόμενη θα είναι στις Βρυξέλλες. τον Οκτώβριο. Και είναι χρήσιμο να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες mm. γιατί ο ρόλος της Κοζάκ κάπως άλλαξε θα έξιζε να ξαναδιαβάσουμε το πρωτόκολλο 1 στο άρθρο 10 αναφέρεται στην Κοζάκ και τις δίνει αρμοδιότητες ευρείας. Εγώ έχω πάει μόνο στη Στοχόλμη και στη Μαδρίτη. Μόνο το να μελετηθεί μόνο ένα σημείο όπως έγινε στο Κόλμη. Δηλαδή με δείγμα πώς λειτουργεί το σύστημα ελέγχου της επικορικότητας δεν ισχύει πια. Διότι η Λισαβόνα προβλέπει γενικό έλεγχο, γενικευμένο έλεγχο της επικορικότητας. Ποιος είναι λοιπόν ο νέος ρόλος με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ δεν θα μιλήσω άλλος. Σωστό είναι να ακούσουμε τον συνάδελφο Μαρτίνες που έχει μακρά εμπειρία του θέματος. και για την τελευταία συνεδρίαση της Κοζάκ και για την επόμενη. Και για το μέλλον της Κοζάκ, ποια είναι η γνώμη που θα μας πει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους. Μην ανησυχείτε. Εμένα με ενδιαφέρε τόσο πολύ το κομμάτι της συζήτησης που άκουσα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Τα προβλήματα που έχουμε, βλέπετε, δεν τα εξηγούμε αρκετά μερικές φορές στα άρθρα που γράφω, αυτή τη βδομάδα γράφω ένα ολόκληρο άρθρο για την πρωτοβουλία πολιτών. Πολλές φορές συζητάμε κλεισμένοι εδώ χωρίς να προβάλλουμε προς τα έξω τις πρωτοβουλίες μας και τις ιδέες μας. Οπότε βρήκα πάρα πολύ χρήσιμη τη συζήτηση αυτή, το ότι άκουσα δηλαδή τους συναδέρφους. Τώρα ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την πρόσκλησή της και για τη δυνατότητα που μου δίνει να έρθω και να σας παρουσιάσω τις εξελίξεις όσον αφορά τις σχέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα σας εξηγήσω ποιες είναι οι εξελίξεις στην ΚΟΖΑΚ. Εδώ θέλω καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μας από την στενή συνεργασία που έχουμε με τον πρόεδρο Καζίνη. Ειλικρινά είμαστε σε μια διαδικασία συμβίωσης που ποτέ ξανά δεν είχαμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως δυσκολία. Όλα είναι εύκολα και μας προκαλούν ικανοποίηση. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν, έχουμε κερδίσει έδαφος από τη στιγμή που ο πρόεδρος τεγματικών υποθέσεων και το Προεδρείο και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου τα βρίσκουν μεταξύ τους τόσο καλά. Με τον Πρόεδρο Καζίνη, εξάλλου, θα συμπροεδρεύσουμε αντιπροσωπεία έξι ευρωβουλευτών που θα πάει στην Ολομέλεια της ΚΟΣΑΚ 24 με 27 Οκτωβρίου. Εκεί θα είναι και ο κύριος Μεσασμίθ που βλέπω εδώ και ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ και η κυρία Μπέρες και ένας από το ΕΛΚ που θα οριστεί. Δεν έχει οριστεί ακόμα, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Πρόκειται για μια σημαντική συνεδρίαση. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τα δύο σώματα του Βελγικού Κοινοβουλίου, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάει πολύ καλά να έχετε υπόψη σας ότι στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν προσωπικότητες όπως είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, του Συμβουλίου, δηλαδή ο κύριος Μπαρόσο, ο κύριος Φαν Ρόμπαλ Και υπάρχουν τρία σημεία στην ημερήσια διάταξη, δύο από τα οποία έχουν να κάνουν άμεσα με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικά Κοινοβούλια. Τι προπτικές δηλαδή για τη σχέση αυτή ανοίγει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μιλάμε επίσης για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ. Και θα συζητήσουμε επίσης και για τον μελλοντικό ρόλο της ΚΟΣΕΚ βάσει της νέας νομικής και πολιτικής βάσης που έχουμε τώρα που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που επίσης είναι σημαντικό αν και δεν μας αφορά τόσο άμεσα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν να πούν τα εθνικά κοινοβούλια γι' αυτό. Το πρώτο θέμα λοιπόν, κοινοβουλευτικός έλεγχος στην ε, ΕΠΑ. Ευρωπαϊκή πολιτική δηλαδή ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχουν διάφορα εθνικά κοινοβούλια, λίγο πολύ δικαιολογημένα, εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες που θα έχει η εξαφάνιση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δικοευρωπαϊκής Ένωσης που ζήτησε βέβαια να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση της ΚΟΣΑΚ. Και εμείς και ο πρόεδρος και εγώ λέμε δεν ξέρουμε αν ζει ακόμα η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λογικό κάποιος εκπρόσωπος να έρθει, αν έχει ήδη πεθάνει, αν έχει ήδη αποδημήσει, εις κύριον τι νόημα έχει. Πολλοί ήμασταν πριν εκεί, τώρα είμαι εδώ. Εμένα προσωπικά δεν θα με ενοχλήσει να έρθει κάποιος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Δικοευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΤΕΟΣ ε, κοινοβουλευτική Συνέλευση της Δικοευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Θέας Δικοευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, είναι αλήθεια ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια αναρωτιούνται κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να τους απορροφήσει και να τους βάλει στο περιθώριο όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι μια τέτοια ανησυχία δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ακριβώς επειδή υπάρχουν οι συνθήκες και επειδή εξαφανίζεται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα ζωντανό θέμα. Ένα θέμα που πρέπει να το συζητάμε χωρίς προκαταλήψεις. Και πρέπει να συμφωνήσουμε τελικά. Άρα χρειάζεται προετοιμασία, υπευθυνότητα και τις καλύτερες δυνατόν προθέσεις από όλες τις πλευρές. Μιλήσατε με τα εθνικά κοινοβούλια και πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο για να προετοιμαστεί η συνεδρίαση αυτή της ΚΟΣΑΚ που αναφέρεται στα τρία θέματα αυτά της ημερήσιας διάταξης. Τα δύο από τα οποία, όπως είπαμε, έχουν άμεση σχέση με μας, που είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο τη ΕΠΑ και το μέλλον της ΚΟΖΑΚ. Οι απαντήσει αναλύονται αυτή την εποχή και καταδεικνύουν μεγάλες διαφορές, για να το πω διπλωματικά και απλά, Διαπιστώνεται δηλαδή δίσταση απόψεων μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ακόμα και μεταξύ δύο ε, βουλών στο ίδιο κοινοβούλιο, δύο σωμάτων δηλαδή μέσα στο ίδιο κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για 27 τελικά σώματα, πρόκειται για 30 τόσα σώματα. Μερικές φορές διαπιστώνονται λοιπόν τεράστιες διαφορές, ακόμα και μεταξύ σωμάτων από την ίδια χώρα. Οι προτάσεις που γίνονται επίσης διαφέρουν μεταξύ τους. Σχετικά με την ΚΟΣΑΚ, δηλαδή πώς θα είναι οι αντιπροσωπείες, ε, πόσα μέλη θα έχουν, πώς θα πρέπει να γίνεται η χρηματοδότησή τους, ε, με τι ρυθμούς θα συνεδριάζουν. Σε όλα αυτά διαπιστώνουμε διαφορές. Μία πάντως από τις επιλογές που διαφαίνονται είναι τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και της κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, σε ποιον θα πρέπει να ανατεθεί η υπευθυνότητα αυτή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η ίδια η Κοζάκ που να το αναλάβει αυτό. Αλλά με αυτή τη θέση συμφωνούν οι λιγότεροι οι λιγότεροι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι δεν έχουν συγκεντρωθεί και συζητήσουν. Ίσως όταν βρεθούμε και συζητήσουμε και ακουστεί η επιχειρηματολογία των ΜΕ και των ΔΕ, να υπάρξουν περισσότεροι πέρα αυτής της ιδέας. Εξάλλου ορισμένα κοινοβούλια δεν έχουν καν αποφανθεί για το θέμα αυτό. Όταν εμείς πάμε σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις, μεταφέρουμε την άποψη του κοινοβουλίου μας. Πολλές φορές όμως τα εθνικά κοινοβούλια μεταφέρουν την άποψη συγκεκριμένων οργάνων ή την άποψη ορισμένων μόνο εθνικών βουλευτών που παρακολουθούν το θέμα και έχουν μια σοφή ίσως άποψη, αλλά χωρίς προηγουμένως να την έχουν συζητήσει με όλους τους υπόλοιπους στη χώρα τους. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την άποψη όλων των κοινοβουλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, έδωσε τις απαντήσεις του. Είναι ε, απαντήσεις που έχει επικυρώσει το Διευρυμένο Προεδρείο των ε, Επιτροπών που ασχολούνται με θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, βάσει των νέων αρμοδιοτήτων και των νέων διατάξεων της συνθήκης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα δομή. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνονται κοινοβουλευτικές συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων και κάποια θέματα ευαίσθητα που έχουν να κάνουν με τον αριθμό των αντιπροσωπιών ή των μελών αντιπροσωπείας των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτά είναι θέματα που μπορούμε να συζητάμε μαζί τους και να καταλήγουμε σε συμφωνία. Ο κύριος Μπρόκ ήταν πολύ επικοδομητικός με τις δικές του προτάσεις και την προηγούμενη εβδομάδα ε, οργανώθηκε από την ε, ΑΦΕΤ και την ΣΕΔΕ μία συνεδρίαση από κοινού με τους εθνικούς βουλευτές. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να αναλύσουμε τις αρμοδιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ, ώστε να εντοπίσουμε δημοκρατικά κενά ή ελλείμματα, για το οποίο ο Μπροκ δεν λέει ότι ναι υπάρχουν, είναι σημαντικό πάντως στη συζήτηση αυτή να προσπαθήσουμε να καθησυχάσουμε λίγο τα πνεύματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν εντάσεις στη συνεδρίαση της Κοζάκη στη Μαδρίτη. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το κείμενο. Το άρθρο του πρωτοκόλου λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια από κοινού αποφασίζουν για την οργάνωση και την πρόθεση της δικαινοβουλευτική συνεργασία ώστε να είναι αποτελεσματική και τακτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Με το πνεύμα αυτό λοιπόν η αντιπροσωπεία μας πρέπει να ετοιμάσει την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ερωτήσεις της Βελγικής Προεδρίας και να δώσουμε την απάντησή μας αυτή τη βδομάδα. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας, και εδώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Εμένα δεν με απασχολεί το να μην είμαστε πολύ άριθμοι, γιατί μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ σημαντικό παρελθόν. Για μένα το ότι έχουμε τον Μέντες Δεβίγο ή τον Νταφ εδώ σήμερα μαζί μας, αυτό και ο πρόεδρος Καζίνη και εγώ είμαστε εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε, υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες αυτό φτάνει. Για το μέλλον, οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια έχει να κάνει και με το ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να αποφασίσουν για τις δικές τους τις θέσεις σχετικά με ένα όργανο, ένα όργανο δηλαδή όπου τα Εθνικά Κοινοβούλια να έρχονται αφού έχουν συζητήσει και εγκρίνει μεταξύ τους τις θέσεις τους. Εμείς αυτό το έχουμε. Ήδη. Φτάνουμε εμείς. Ενώ από την άλλη μεριά δεν προηγείται αυτή δεν υπάρχει αυτό το όργανο στο οποίο θα καταλήξουν τα εθνικά κοινοβούλια έχοντας πάρει τις αποφάσεις τους. Χρειάζεται λοιπόν το όργανο αυτό. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να έχουμε 47 διαφορετικά σώματα και από την άλλη μεριά ένα. Στις τελευταίες συνεδριάσεις της ΚΟΣΑΚ είδαμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια χρειάζονται ένα συντονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Μαδρίτη, αλλά και εδώ, στις Βρυξέλλες, ποιος θα έρθει. Ο Φάνο Ρομπάλ και ο Μπαρόσο. Και θα μιλήσουν στα εθνικά κοινοβούλια. Κανονικά έτσι είναι δεν θα απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτική βάση έχουν επαφή. Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπείται με μία θέση σχετικά με την οποία έρχεται Κάποιο, ο ο Ρομπά, ο οποίος μιλάει σε 20 τόσα κοινοβούλια ή σε 40 τόσα σώματα και επαναλαμβάνει για τον καθένα του τα ίδια. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτάνει μαζί, Ω ένα σώμα. Χωρίς να ψηφίζουμε ή να αποφασίζουμε με κάποια τέτοια διαδικασία εδώ τις αποφάσεις της ΚΟΖΑΚ. Οι αποφάσεις αυτές έχουν κάποια ρητορική ίσως αξία. Αλλά δεν πειράζει. Όταν γίνουν πολιτικές όμως αποφάσεις, προσοχή. Γιατί η εντύπωση που σχηματίζει κανείς είναι ότι φτάνει να υπάρχουν δύο ή τρία εθνικά κοινοβούλια που να έχουν διαφορετική άποψη σαν να θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους οι υπόλοιποι, σιωπούν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά περιορίζει τη δικιά του τη θέση για να ε, μικρύνει τη ζημιά και τελικά το έγγραφο το οποίο αποφασίζεται είναι έγγραφο το οποίο υπογράφει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά που να μην λέει πράγματα με τα οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει το κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, το κοινοβούλιο μα δεν μπορεί να αποφασίσει. Μπορεί τα εθνικά κοινοβούλια να το βρίσκουν καλό, ναι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω όμω, για παράδειγμα. Το θεσμικό έγγραφο που συζητάμε και υπογράφεται απειλεί τη δημοκρατία, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει τις αρμοδιότητες του. Ο εκδημοκρατισμός της διαδικασίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος τα τελευταία 50 χρόνια βασίστηκε στις όλο αυξανόμενες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που να πιστεύουν ότι αν εμείς αυξάνουμε τις δυνατότητες ελέγχου που έχουμε απέναντι στο Συμβούλιο, που όντω αυξάνουμε αυτές τις δυνατότητες, εννοείται, αν έχουμε συναπόφαση τώρα σε ένα τεράστιο χώρο, ενώ πριν είχαμε σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, ε, προφανώς και έχουμε κερδίσει πολύ όσον αφορά τις αρμοδιότητές μας. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που πιστεύουν ότι αυτό περιορίζει την δημοκρατία στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Γιατί τα εθνικά κοινοβούλια πιστεύανε μέχρι τώρα ότι έχουν το μονοπόλιο ελέγχου του Συμβουλίου, το οποίο είναι λάθος. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις κυβερνήσεις τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτή είναι μια αρμοδιότητα και μια δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπετε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητάμε μαζί τους. μια συγκεκριμένη θέση του ενός ή του άλλου κοινοβουλίου λέμε είναι η μειοψηφία. Ναι, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή η μειοψηφική θέση όταν τίθεται και τίθεται έτσι έντονα έχει σαν αποτέλεσμα τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια να σιωπούν. Και ναι, με στους διαδρόμους σου λένε μπα, δεν, δεν νομίζω κτλ. Ναι, αλλά στην Ολομέλεια δεν λένε τίποτα. Και άρα προχωράει αυτή η μειοψηφική άποψη. Και εμείς αναγκαζόμαστε να χαμηλώσουμε τους τόνους. Σε ένα βαθμό βέβαια. Δεν λέω ότι θα τελείως, αλλά είναι σε αντίφαση με αυτά τα οποία έχουμε καταλήξει εμείς. Και τελικά το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα με το οποίο δεν συμφωνεί και τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και στο μέλλον να χρησιμοποιούμε τη σημερινή ΚΟΖΑΚ Πολύ ωραία να τη χρησιμοποιούμε. Εννοείται είναι ένα σώμα που δουλεύει. Δεν χρειάζεται να είναι το μόνο, μπορεί να συμπληρωθεί από άλλα. Αλλά, όπως και να έχει το πράγμα, λέω, Καζίνη, ότι λείπει μία μονάδα που να συντονίζει τα εθνικά κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετέχει, να μην συμμετέχει, να είναι παρατηρητής μόνο. Αλλά δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφίσταται αυτά τα οποία ε, αποφασίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια αν δεν τα αποφασίζουν με πλήρη νομιμότητα. Δεν μπορεί το, τα Εθνικά Κοινοβούλια να πατάνε τον γκάζι και εμεί το φρένο. Δεν γίνεται. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Υπάρχει θέληση, υπάρχει πρόθεση να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα βγει από τη συνεδρίαση των Βρυξελών πρώτα. Είναι πολύ καλά οργανωμένη όσον αφορά τις υποδομές, την τεκμηρίωση και προεδρεύει πολύ αποτελεσματικά, προεδρεύεται πολύ αποτελεσματικά και πιστεύω ότι πρέπει να συγχαρούμε της υπηρεσίας μας, της Γενικής Διεύθυνσης και κυρίως την Κριστίν Βερζέ, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη δουλειά αυτή. Αυτά είχα να σας πω. Ήρθα εδώ για να ακούσω και εσάς, για να μάθω από τις εμπειρίες των συναδέρφων που είναι εδώ παρόντες. Και επίσης, σας ζητώ να συνεχίσετε να δουλεύετε και με τον Καζίνη και με μένα. Να ξέρετε ότι αυτό που δεν θα γίνει, το βέβαιο είναι, το τελευταίο που θα γίνει δηλαδή, είναι να μην συνεργαζόμαστε εμείς καλά. Αποκλείεται. Γιατί ο πρόεδρος Καζίνη και εγώ συνεργαζόμαστε τέλεια, οπότε και η συνεργασία γενικότερα μεταξύ μας θα πάει πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Σύμφωνα κι εγώ ότι μέχρι στιγμή μεταξύ μας δεν υπήρξε σύγκρουση και ελπίζω να μην υπάρξει. Επιτρέψτε μου πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να πω δύο λόγια αυτό που είπα πριν και ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου. πρέπει να οριστούν οι μελλοντικέ αρμοδιότητες της ΚΟΖΑΚ με βάση το άρθρο 10 του περίφημου πρωτοκόλλου υπαριθμών 1. Δεδομένο είναι δύο πράγματα είναι δεδομένα. Πρώτον, δεν έχει σημασία να υποβάλλονται στην ΚΟΖΑΚ επιμέρους ερωτήσεις, ή νομι... επιμέρους νομοθετήματα του Κοινοβουλίου, νομοθετικές προτάσεις Αυτό μπορεί να γίνεται με άμεση επαφή με τις επιτροπές ή με την Κομισιόν, συγγνώμη. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν δεν υπάρχει. Δεύτερον, έχεις δίκιο όταν λες ότι είναι μια συνεδρία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εμείς, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, εμείς είμαστε μία από 40 περίπου. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει ένας ε, χαρακτήρας ξένου σώματος κατά κάποιο τρόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πλειοψηφία των εθνικών αντιπροσωπιών είναι αυτή που είναι. Αν δούμε όμως πιο βαθιά ποιος είναι ο ρόλος της ΚΟΖΑΚ δεν είναι για να γίνουν προτάσεις προς το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, του Συμβούλιο για συγκεκριμένα θέματα και μέτρα. Όχι, είναι ένας τρόπος να καταγράφονται κάθε φορά να καταγράφεται η κατάσταση των πραγμάτων. Μερικές φορές μπορεί να συζητώνται θέματα πιο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά. Αυτό δικαιολογεί και καθιστά μάλλον αναγκαία την παρουσία της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου. Παράδειγμα, συζητάμε το ενιαίο εκλογικό νόμο που έχει σχέση με την ιδέα που έχουμε για την Ευρώπη. Είναι ένα επιμέρους μέτρο, μεν, αλλά αφορά σε βάθος τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό μπορεί να συζητηθεί στην ΚΟΖΑΚ. Θα μπορούσε να προταθεί στην επόμενη συνάντηση την τριμερή. Το δίνω ως παράδειγμα. Ο μελλοντικό ρόλο λοιπόν της ΚΟΖΑΚ μπορεί να ενισχυθεί στο μέλλον. Τα εθνικά κοινοβούλια μέσω των ειδικών επιτροπών τους, που ασχολούνται με την Ένωση ενώ, να συζητάνε όχι μόνο το πώς θα γίνεται ο επιμερισμός των διαρθρωτικών κονδυλίων κλπ, αλλά και για πιο σοβαρά θέματα. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο συνάδελφος Νταφ. κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ε, Μιγγέλ Μαρτίνες για την πολύ επιδέξια παρουσίαση σύνοψη της σημερινής κατάστασης. Στην Κοζάκα. Η συνθήκη λέει ότι οποιοδήποτε νέα αρρύθμιση θα πρέπει να αποφασίζεται από κοινού μεταξύ ημών και των εθνικών κοινοβουλίων. Δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους στα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό, στη συνάντηση των Βρυξελών, θα πρέπει ευγενικά μεν, αλλά στεναρά, να τεθεί το σημείο αυτό. Η συνθήκη επίσης λέει ότι πρέπει να φροντίσουμε να βελτιωθεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μερικοί συνάδελφοι θεωρούν ότι αρκεί το status quo και ας εφησυχάσουμε για το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση και να στρατολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια, να τους βοηθάμε, να τους συμβουλεύουμε, να ζητάμε τη γνώμη τους πολύ περισσότερο από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Θα αναφερθώ μόνο στην θέμα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. γιατί το διευρεμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα το θέμα αυτό. Ε, με θέμα αυτό. Θα βοηθούσε πολύ αν ο κύριος Μαρτίνες μπορεί να είναι παρόν. Θα ήταν μια σημαντική συνέχεια ως προς τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχουν τρία διαφορετικά θέματα. Για τα Εθνικά Κοινοβούλια σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Τρία πράγματα προπέπει να έχουν διακριτές αρμοδιότητες. Είναι θέματα που αφορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια, είναι θέματα που αφορούν το Ευρωκοινοβούλιο, προπολογισμό, ορισμός στην ε, διορισμή στην υπηρεσία εξωτερική δράση κλπ. Αυτό είναι δικό μα ρόλο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και θα πρέπει να προστατεύσουμε το ρόλο αυτό από τυχόν εισβολέ εκ μέρου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο στοιχείο η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. όπου χρειάζεται κοινή προσπάθεια μεταξύ ημών, ήτα και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να καθοδηγήσει την συζήτηση προς το τρίτο αυτό σημείο, ως προς το τρίτο σημείο, να αποφευχθεί σύγχυση και τυχόν ζηλοτυπία. Του να θέλει ο καθένας να τραβήξει τη κουβέρτα προ τη δική του μεριά. Επίσης πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το ρόλο της κοζάκη και θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αυτό για μας είναι παράδεκτο. που αντιπροσωπεύει την εξουσία του κοινοβουλίου μας κάτι τέτοιο. Ναι, να έχουμε κοινέ συνεδριάσεις και μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών επίσης κοινέ συνεδριάσεις, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει σε μία αντιπροσωπεία με 35-40 μέλη τότε θα μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό διάλογο για ουσιώδη θέματα πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αλλάξει την ιστορική του λειτουργία. Πρέπει να ορίσει μια αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την ΣΕΝΤΕ που θα συνεδάζει σε αυτή την κοινή επιτροπή. Δεν θα το πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό όποιος θέλει να έρχεται όποτε θέλει. Γιατί αν το επιτρέψουμε αυτό, δεν θα έρχονται τα οι βουλευτές θα βρίσκουν άλλα πράγματα να κάνουν. Θα πρέπει να υπάρχει επίσημα μια αντιπροσωπεία κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών τη ειδικών για θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Όχι μια νέα επιπλέον γραμματεία, Έχουμε τους υπαλλήλους που χρειαζόμαστε. Αρκούν. Απλώς χρειάζεται να αναβαθμιστεί η ουσία της δουλειάς που κάνουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Μέντες Δεβίγκο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Μαρτίνες. Ακούγοντάς τον, θυμόμουν κάποια άλλη περίπτωση με τον Ιμπένι στην Κοζάκ και την κυρία Φοντένα, άλλο δίδυμο εκεί, που πριν από 15 χρόνια λέγανε το ίδιο που λέτε κι εσείς τώρα, ότι δηλαδή το πρόβλημα της Κοζάκ είναι ότι δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει με την Κοζάκ, όπως έλεγε και ένας ε, φιλόσοφος από την Μαδρίτη. Εμείς όμως φτιάξαμε την Κοζάκ και εμείς είμαστε ιδρυτές της Κοζάκ και εξακολουθούμε να είμαστε μέσα στην Κοζάκ. Μπορεί κανείς ε, να μπει στον πειρασμό να πει «Μπα, αφού έχει γίνει αδύνατη η ζωή μας εκεί μέσα, να την εγκαταλείψουμε». Ε, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο ώστε η Κοζάκ να παίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Κοζάκ δεν είναι τα εθνικά κοινοβούλια. Όχι. Είναι ειδικέ επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων. Δηλαδή, οι βουλευτές που πάνε, και το είπατε και εσείς πολύ καλά στην Κοζάκ, δεν εκπροσωπούν τα εθνικά κοινοβούλια. Εκπροσωπούν ούτε καν το σώμα τους. Είναι ενδιαφέρον, αλλά πρόκειται για συγκεκριμένες ειδικέ επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για να μιλήσουμε, για να ενημερωθούμε. Ναι, καλές είναι αυτές οι ειδικέ επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά τα κοινοβούλια στο σύνολό τους, και εγώ έχοντας μιλήσει με διάφορου εθνικού βουλευτέ το ξέρω, στο σύνολό του δεν εκπροσωπούνται εκεί. Αυτό το όνομα ΚΟΖΑΚ είναι ειδικέ επιτροπές σε κοινοτικά θέματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τίποτα άλλο. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι μια που είναι χρήσιμο υπάρχει και στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας αλλά θα κάνουμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το όργανο αυτό. Και πώς. Πρέπει να ετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά και να ετοιμαστεί πάρα πολύ καλά η Τρόικα. Είναι κεφαλιόδους σημασίας. Να χρησιμοποιήσουμε την Τρόικα λοιπόν. Ο κ. Μαρτίνες έχει δίκιο. Τον τελευταίο καιρό είμαστε λίγο στην αμυντική θέση στην Τρόικα. Ο πρόεδρος Καζίνη είπε κάτι ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα συζητήσουμε την έκθεση DAF για μια τροποποίηση της πράξης του 96. Ωραία, γιατί να μην το θέσουμε αυτό εκεί και τα Εθνικά Κοινοβούλια ή οι ειδικέ επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων να μας πούν τη γνώμη τους. Δηλαδή, μην περιμένουμε κάθε φορά να δούμε αυτοί με τι θα έρθουν, να πηγαίνουμε και εμείς εκεί με θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε σημαντικά. Να ετοιμάζουμε λοιπόν την Τρόικα. Δεύτερον, Σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, είναι στην ημερήσια διάταξη τώρα, αλλά την εποχή του Ιμπένη και της Φοντέν δεν ήταν. Ήταν επικουρικότητα. Κάποια στιγμή κατάλαβαν τα εθνικά κοινοβούλια ότι εμείς δεν παρεβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας σε συστηματική βάση. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε και πριν, είναι κοινότητα δικαίου. Άρα τηρούνται οι αρμοδιότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών. Και αυτό ισχύει και στην εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Τώρα με κάθε σεβασμό και μάλιστα σε κάποιον που συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να ελέγξει την εξωτερική πολιτική του οποιοδήποτε το όργανο αυτό. Ποτέ. Τίποτα δεν έλεγχε. Εν το επιχείρημα που λέει ότι αφού η συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης εξαφανίστηκε, ας φτιάξουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν συμφωνώ. Να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Και πάλι με κάθε ειλικρίνεια Ούτε πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι όπως λέμε ότι είναι θέματα για πρίγκιπες και όχι για την πλέμπα. Ε, και εδώ είναι θέμα που οι κυβερνήσει κρατάνε στα χέρια του. Φυσικά και λογοδοτούν και έρχονται και μα λένε και τα λοιπά. Και η συνθήκη τη Λισαβόνα μα έκανε να προχωρήσουμε πολύ. Είναι υποχρεωμένοι να έρχονται και να μα λένε. Πριν ερχόσα δύο φορέ το χρόνο, μα ακούγανε και χαίρετε αντίο σα. Τώρα είναι κάτι παραπάνω. Ελέγχουμε κάπω την εξωτερική πολιτική, ναι, αλλά μην υπερβάλλουμε. Σε ένα βαθμό μόνο. Κατά τα άλλα πιστεύω και συμφωνώ με τον Άντριου Νταφ για το ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νέα όργανα για τέτοια πράγματα. Και υπενθυμίζω ότι υπήρξε στην κοινοβουλευτική συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης υπήρχε μια ιδέα που την ήθελε ο Ζισκάρδεστα ο πρόεδρος τότε για το Κογκρέσο των Λαών. Αλλά τελικά καταλήξαμε στο ότι δεν ήταν κάτι καλό. Αφού δεν υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας, τώρα τι κάνουμε, ψάχνουμε έναν άλλο τρόπο για να το δημιουργήσουμε και πάλι. Όχι. Ούτε τότε μου φαινόταν καλή ιδέα, ούτε σήμερα. Τον εισαγάγουμε συγκεκριμένα θέματα, γιατί η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι κάτι αφηρημένο. Χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα όταν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Το να κάνουμε προσκλήσεις επιμονή μου βάσεως στις επιτροπές όχι των κοινωνικών κοινοτικών θεμάτων που πάνε έτσι και αλλιώς στην ΚΟΣΑΚ, αλλά εξωτερικών υποθέσεων, για παράδειγμα, των Εθνικών Κοινοβουλίων, πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό. Να έρχονται και να συμμετέχουν στι συνεδριάσει μα. Εμεί είμαστε πιο γενναιοδοροί από πολλά εθνικά κοινοβούλια που δεν μα αφήνουν εμά να ε, πηγαίνουμε στι δικέ του συνεδριάσεις, έστω ω παρατηρητέ. Όχι, εγώ λέω εκείνοι να έρχονται και να συμμετέχουν. Βεβαίω, ευχαρίστω να έρθουν, να παρεμβαίνουν, να συζητάνε, γιατί όχι. Να το ζητήσουμε αυτό. Και κάτι άλλο που χρησιμοποιούμε, αλλά ίσως πρέπει να δώσουμε μια καλύτερη μορφή. Εκείνες οι Joint Parliamentary Meetings, όπως τις λέμε. Τρεις το χρόνο, δύο το χρόνο κάνουμε, να αφιερώσουμε ένα μέρος τους και σε αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να παίξουμε έξυπνα και να βγούμε από το αδιέξοδο Βάζοντα με διαφορετικό τρόπο να συμμετέχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια στα κοινοτικά ζητήματα. Τώρα κάτι άλλο που μπορεί να μην είναι πολύ σεξι, αλλά τι να κάνουμε. Και φοβάμαι ότι ο αντιπρόεδρο Μαρτίνες πρέπει να βρει τρόπο να το περάσει. Θυμάμαι, ήταν επί Βρετανικής Προεδρίας. Θα το θυμάται και Είχαμε την Κοσάκ στο Λονδίνο. Και ο κύριος Πρέσκοτ δεν του είχαν πει ότι εκτός από τα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν εκεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 30 λεπτά λοιπόν μίλαγε και έλεγε τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα Εθνικά Κοινοβούλια και ξανά τα Εθνικά Κοινοβούλια. 30 λεπτά μετά σηκώθηκα και του είπα «Ξέρετε, κάτι σας έχει λείψει εδώ». Και εσείς έχετε χιούμορ κύριε Μαρτίνεθ. Χρειάζεται βοήθεια μερικές φορές από διάφορες πλευρές για να βγούμε από αδιέξοδα. Ο ίδιος φιλόσοφος που σας έλεγα και πριν από τη Μαδρίτη έλεγε για την Ισπανία ότι πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε. Ε, λοιπόν, και εμείς εδώ πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε. Ας φροντίσουμε λοιπόν να συνεπάρχουμε. με χιούμορ και με υπομονή όπως είχε και ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Eh, eh, eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, συνάδελφο Μαρτίνες για τις πληροφορίες που μας έδωσε και για τα θετικά της ΚΟΖΑΚ. Εγώ θα επικεντρωθώ στο θέμα το οποίο περισσότερο ακούστηκε και από τη δικιά σας παρέμβαση και από τους συναδέλφους. Το θέμα της ασφάλειας και άμυνας. Κάποια στιγμή είπατε δεν έχει σημασία ποιος κάνει τι. Το θέμα είναι να γίνεται και να γίνεται καλά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Εθνικό Κοινοβούλιο να γίνει πριν, τώρα, μετά. Αν το τι έκανε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι τελικά κανείς δεν το κάνει. Και ότι υπάρχει ένας μεγάλος χώρος με κενά. Άκουσα τον ε, κύριο Μέντες Βίγο που είναι συνταγματολόγος και σωστά τα λέει. Στη δημοκρατία Τίποτα σημαντικό που έρχεται από και έχει να κάνει με τους πολίτες δεν πρέπει να μένει εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα σημαντικά. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν. Οι κυβερνήσει μπορεί να έρχονται να εξηγούν περισσότερο λιγότερο, αλλά υπάρχει υποχρέωση. Είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα δεν γίνεται. Ούτε τα εθνικά κοινοβούλια κάνουν τον έλεγχο αυτό, ούτε κανένα άλλος. Ήμουν βουλευτής στη χώρα μου. Η άμυνα δεν είναι το ίδιο με την ασφάλεια. Άμυνα σημαίνει εξοπλισμός, στρατιωτικό σκέλος. Και η ασφάλεια που ελέγχουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι η εθνική, δεν είναι η ευρωπαϊκή η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία επίσης ήμουν μέλος, όντω είναι ένα μετριοπαθή οργανισμός. Θα συμφωνήσει όμω ο κύριος Μαρτίνεθ ότι η ποιότητα των εκθέσεών τη μας εξέπλητε όλους. Με λίγους τεχνικούς και υπαλλήλου κατάφερνε να καταλήγει σε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Υπάρχουν μπορείτε να τις δείτε σε βάθος εκθέσεις που δεν έχουν γίνει ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα, ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εγώ έχω συμμετάσχει και στα τρία όργανα. Τέλος. Πρέπει να προσπαθήσουμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και κυρίως την Υποπιτροπή της ε, ΣΕΔΕ, που είμαι εγώ μέλος, να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες πρωτοβουλίας, ώστε τα Εθνικά Κοινοβούλια να συντονίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον έλεγχο της κοινή ασφάλειας, η οποία και προσοχή, πολλές φορές έχω πει προσοχή, ούτε και αυτήν την ελέγχουν οι διάφορες αποστολές για την ειρήνη. Ο συμπατριώτης μου Σολάνα έκανε μεγάλη δουλειά, αλλά να ξέρετε ότι κάθε φορά περιοριζόταν νομικά και δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα. 20 ειρηνευτικές αποστολές λοιπόν και πρόθεσης της ειρήνης παραδειγματικές έγιναν. Αλλά δεν είναι αυτές οι αποστολές που κάνουν την ασφάλεια στην Ευρώπη. Έχει και άλλα στοιχεία. Πολιτικά, πολιτιστικά, δημογραφικά, τρομοκρατία, διεθνές έγκλημα. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ή ε, κάθετος και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να φροντίζουν για αυτή πολύ πιο οργανωμένα από ό,τι το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δύο λόγια έχω να πω. Πρώτον, επιτέλους, το Δεκέμβριο εξαφανίζεται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρω εγώ, επίσημα πάβει τις δραστηριότητές της, ιδέω. Προσοχή όμως. Τι την αντικαθιστά. Γιατί έχει, είχε μεγαλύτερη κυβερνητική διάσταση. πρέπει να αναλάβουν τις αρμοδιότητες αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά προσοχή πώς θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από αυτά που συζητάμε εδώ είναι υπομονή και προσοχή, σοφροσύνη. Να είμαστε παρόντες, αλλά προσοχή σε δύο άξονες. Πρώτον, δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε ότι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Συμβουλίου και των κυβερνήσεων τον κάνουμε εμείς και δεύτερον δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς μια διαδικασία συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια γιατί υπάρχει η επικουρικότητα που έχει το δικό της δρόμο, υπάρχει το steering group μέσα στο οποίο δουλέψαμε για τη δημιουργία ενός πλαισίου σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου προβλέπονται διάφοροι μηχανισμοί. Αυτόν τον άξονα να ενισχύσουμε, αυτή τη διάσταση. Γιατί εμείς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε έναν άξονα για το συντονισμό των εργασιών μας. Υπομονή και σοφροσύνη λοιπόν. Ο κύριος Μαρτίν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους, που όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και επικοδομητικά, ανοείται. Ο κύριος Άντριου Νταφ βγήκε, αλλά θέλω να το απαντήσω. Ας σημειώσει κάποιος. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει, για το ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις. Γιατί η συνθήκη πραγματικά καθορίζει ένα νέο επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού. Σωστά και υπάρχει ένα πρώτο βασικό στοιχείο, το είπε ότι χρειάζεται ορθολογισμός. Πιστεύω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια εξορθολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πέντε συνεδριάσεις επιτροπών μέσα σε ένα μήνα και τον επόμενο να μην γίνει καμία, οι άλλες επιτροπές να συνεδριάζουν τρεις φορές και άλλε καθόλου. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόοδο και αποτελεσματικότητα. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Σιγά σιγά, με υπομονή. Τέλεια. Να μην υπάρχει όμως παρεξήγηση εγώ πιστεύω ότι την ΚΟΖΑΚ πρέπει να τη διατηρήσουμε και να αποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από την ύπαρξή της. Μα η συνθήκη προβλέπει τη διατήρησή της, οπότε προφανώς και παραμένει. Έλεγα πριν ότι υπάρχει κάτι αναπόφευκτο νωρίς ή αργά και είναι ένα συντονιστικό όργανο για τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα συζητάει παρουσία ημί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία δομή όπου ισομερός, όχι 47-1 ή 27-1, ισομερός λοιπόν να συγκεντρώνει εκπροσώπηση των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί τελείωσε το πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι 27-47-32 από τη μία και από την άλλη εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα εκθέτουν το πρόβλημά τους, το κοινοβούλιο να εκθέτει το δικό του ζήτημα, τη δικιά του θέση και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Αυτό χρειάζεται. Η ισοτιμία, η ισομερής εκπροσώπηση των δύο πλευρών. Γιατί Κοζάκ, έτσι όπως έχει σήμερα, όσο δεν εγκρίνει έγγραφα, δεν υπάρχει πρόβλημα. 47 ένας, 27 ένας, κανένα πρόβλημα. Όταν όμως εγκρίνει κάποιο έγγραφο, ε, τότε δεν γίνεται. Γιατί τα έγγραφα που εγκρίνονται μπορεί να είναι πολύ στοιχειώδη, πολύ γενικά, αλλά μπορεί να είναι και έγγραφα τα οποία δεσμεύουν με αυτά που λένε. Και εκεί είναι που πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από το διέξοδο. Τι θα πούμε, η Κοζάκ να μην εκπονεί κανένα έγγραφο με συμπεράσματα ή αν υπάρχει ένας που δεν θέλει κάτι δεν πρέπει να μπαίνει μέσα στο έγγραφο ή όπως έγινε στην τελευταία συνεδρίαση όπου τελικά ψηφίζουμε κάθε παράγραφο χωριστά. Εδώ βλέπω δηλαδή μια κατάσταση που δεν είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξαν κείμενα με τα οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν είναι το λιγότερο κακό. Μία παράγραφος που μπορεί να την έχουμε διορθώσει να είναι μια παράγραφος που παραμένει να λέει κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε, ε, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η παράγραφος. Και δεν μπορεί να πρέπει δέκα φορές να σηκωνόμαστε και να πρέπει να λέμε κάθε φορά το ίδιο δεν το θέλουμε. Ε, και εδώ χρειάζεται εξορθολογισμός. Εφόσον η Κοζάκ εγκρίνει έγγραφα είτε συμπεράσματα είτε κάτι άλλο, η έγκριση αυτή πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό όλων των πλευρών. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να ξέρετε επίσης ότι έχουν μεγάλη δύναμη τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εθνικά Κοινοβούλια ή σώματα μερικές φορές έχουν λίγες δραστηριότητες και άρα άπειρο χρόνο για να επεξεργάζονται αυτά τα ζητήματα επιπλέον έχουν σχετική εκπροσώπηση των πολιτών στις χώρες τους. Στην ΚΟΣΑΚ δεν λένε ειδική επιτροπή, λένε τη χώρα. Γαλλία, Λιθουανία, Ισπανία. Οπότε σηκώνονται και δεν λένε εγώ μιλάω εκ μέρους μιας ειδική επιτροπής. Όχι, όχι, όχι. Λένε εκ μέρους της χώρας. Αυτό πρέπει να πετύσουμε να αλλάξει. Αυτά για τον ΤΑΦ. Επίσης και εγώ είμαι πεπισμένο ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο σώμα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τη ασφάλεια και άμυνα, όπως το έχουν πει και κάποια εθνικά κοινοβούλια. Δεν θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε αυτό. Αυτό όμω, που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Δηλαδή αυτά που έγιναν 15 χρόνια, τα λέω αυτά στον ίδιο, δεν είναι τα ίδια με σήμερα. Εσύ τα ξέρει καλύτερα από μένα. Τώρα έχουμε διαφορετική νομική βάση, με διαφορετική συνθήκη και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση. Και να ανταποκριθούμε με κοινή λογική βέβαια. Όπως έλεγε και ο Λουίς, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε κορποριστές, δεν είναι αυτό, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο συνεταιριστικά, ούτε με πατριωτισμό. Όχι, είναι θέμα υπευθυνότητα και της καλύτερη αποτελεσματικότητα. Σωστά, Λουίς. Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση δεν ήλεγχε. Με οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό όργανο ελέγχει και προσανατολίζει. Πάντως έχεις δίκιο Λουίς ότι ήταν αποτελεσματική. Αλλά ήταν λιγάκι σαν πανεπιστήμιο, όπου εκεί πηγαίνανε διάφοροι σημαντικοί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνανε ομιλητές. Και ακούγανε τις ερωτήσεις των βουλευτών. Έχεις δίκιο όπως και να έχει το πράγμα, Λουίς, για το ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί. Ο Άντριου κάποια στιγμή είχε πει ότι έπρεπε να υπάρχει μια ειδική αντιπροσωπεία για να μην είναι άλλη τη μια και άλλη την άλλη, να είναι μόνιμη τα μέλη. Δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Και για τον Χαουρεγκή, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούμε να αποσυρθούμε. Δεν συζητιέται αυτό. Συζητιέται το αν εγκρίνονται ψηφίσματα και πώς εγκρίνονται. Αυτό ναι ώστε η τάση, ο πειρασμό που υπάρχει να βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν εχθρό, σαν αντίπαλο, σαν μια υπερελιστική δύναμη, δεν μπορεί αυτό να σκέφτονται άμα δεν θέλουμε να εγκρίνουμε κάτι. Όχι, εγώ. Σε βλέπω ότι διστάζεις. Σου είπα ότι τα κοινοβούλια έχουν την τάση να δείχνουν την αλληλεγγύη τους απέναντι σε κάθε διαφωνούντα μεταξύ τους. Για τους υπαλλήλους τώρα των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι στις Βρυξέλλες. Έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Μεταφέρουν πληροφορίες, ενημερώνουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι και πάλι πρέπει να φροντίσουμε για το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια, να δώσουμε και σε αυτούς έναν πιο σημαντικό ρόλο. Να μην είναι ένα γραφείο χωρίς τίποτα άλλο από το να στέλνει επιστολές. Ο πρόεδρος Κασίνη θα συμφωνήσει σίγουρα μαζί μου για το ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους υπαλλήλου οι οποίοι στις δικές μας πολιτικές ομάδες δουλεύουν πολύ αποτελεσματικά για τον σκοπό μας και κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Πριν αναφέρθηκα στους υπαλλήλου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θέλω να αναφερθώ και στους υπαλλήλου των πολιτικών ομάδων που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να προχωρήσει αυτή η επόθεση και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό να το πω αυτό. Και αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είναι μόνο λόγια. πραγματικά το πιστεύω. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να λέγεται και αυτό. Γιατί εύκολα επικρίνουμε, πρέπει να επικρίνουμε όταν υπάρχει λόγος να επικρίνουμε, αλλά εξίσου εύκολα πρέπει να λέμε και τον μπράβο και να ευχαριστούμε και να αναγνωρίζουμε με τη διπλή έννοια του όρου. Να αναγνωρίζουμε ότι όντω εκτελούν έργο και να αναγνωρίζουμε να του ευχαριστούμε δηλαδή για την καλή του δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Αντιπρόεδρο Μαρτίνε για τα τελικά του αυτά λόγια. Δεν τελειώσαμε όμω, γιατί ακόμα δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Μέντε Δεβίγκο πρώτο. Πολύ σύντομα και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο. Είναι πολύ δύσκολο να μην εγκρίνει συμπεράσματα η Κοζάκ. Πάντα το κάνουμε, θα συνεχίσει να το κάνει. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό που εξηγήσατε, πρέπει να βάλουμε την Τρόικα να δουλέψει πιο πολύ. Δηλαδή να φροντίσουμε ώστε το τελικό έγγραφο να μην έχει τίποτα που μας ενοχλεί. Τώρα αν τελικά υπάρχει κάτι που εσεί, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να ε, συνυπογράψουμε, ε, να μην το κάνουμε. Έχετε δίκιο. Και εγώ αναγκάστηκα να υπογράψω μερικές φορές ξέροντας υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ε, μου αρέσανε και που αντιβαίνανε μερικές φορές και με το κοινωτικό δίκαιο. Αναγκαστήκαμε. Ε, λοιπόν, πρέπει και αν είδε το πρόσωπό μου έτσι κάπως διστακτικό, είναι γιατί πιστεύω ότι θα εξακολουθεί να εκδίδει συμπεράσματα ε, Κοζάκ. Αυτό που δεν βλέπω πολύ ξεκάθαρο είναι το θέμα του συντονισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Όπως έλεγα και πριν, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που αποτελούν μία ενότητα. Και δεν ξέρω αν θα θέλανε να στείλουν μια αντιπροσωπεία τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να εκπροσωπούνται σε ένα συντονιστικό όργανο. Τα εθνικά κοινοβούλια, όχι οι ειδικέ επιτροπές. Η ιδέα μιας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να δουλεύει με ένα συντονιστικό όργανο των Εθνικών Κοινοβουλίων για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής μου φαίνεται περίεργο. Να το ξανασυζητήσουμε αυτό πριν βάλουμε το θέμα επιτάπητος. Thank you very much, President. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν παρακολούθησα όλη τη συζήτηση, αλλά έχω μια καλή συνεργάτη εδώ που θα με πληροφορήσει. Φυσικά και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις, γιατί πρέπει να ανταλλάζουμε απόψει. με τους αντιπρόεδρους που ασχολούνται με συγκεκριμένο θέμα, και δικά μου αυτό. Όλοι ξέρουμε στις τελευταίες εκλογές, στις 42 τις εκλογές, μόνο 42% ψήφισαν. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε εμά και στους Ευρωπαίους πολίτες. Χαίρομαι λοιπόν γιατί ότι το πρωί είχαμε πάρα πολλού συναδέλφου που άκουσαν αυτή τη συζήτηση για την πρωτοβουλία των πολιτών. Βέβαια, εμεί είμαστε υπεύθυνοι να βρεθεί ένα σύστημα καλό για όλους. Πρέπει λοιπόν η παρουσία μας στην Κοζάκ να παραμείνει. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και η Κοζάκ να εξακολουθήσει να είναι ένα φόρουμ για ανταλλαγή εμπειριών χωρίς συγκεκριμένε αρμοδιότητες για το θέμα άμυνας όπως αναφέρθηκε λίγο πιο πριν έχουμε την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση ως τρόπο χειρισμού αυτού του θέματος. Φυσικά χρειαζόμαστε συντονισμό. Όλοι ξέρετε ότι είμαι υπέρ της ισότητας, όχι μόνο ισότητα μεταξύ των φύλων, ισότητα και ισοτιμία και να ξέρουμε ποιος κάνει τι σε κάθε σύστημα. Αν το σύστημα λοιπόν είναι ισομερές, θα έχουμε καλύτερη καθοδήγηση. Ευχαριστώ και εγώ τον Αντιπρόεδρο για το έργο του ως προς την ΚΟΖΑΚ. Τέτοιου είδους συζητήσεις τις χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε πολύ λίγοι οι παρόντες. Έχουμε προβλήματα άλλο γιατί εγώ είχα μια ομάδα επισκεπτών, έπρεπε να απουσιάσω για λίγο. Επαλαμβάνω όμως έχουμε τη γραμματεία η οποία θα μας πληροφορήσει για το τι υπόθηκε και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ομάδα που είναι εδώ στην αίθουσα που προετοίμασε όλες τις συναντήσεις αυτές. Κοινή δουλειά, κοινό έργο, με τη βοήθεια όλων. Πρόεδρος. Τώρα φτάσαμε πραγματικά στο τέλος. Χθες τους συντονιστές επιφορτίστηκε ο αντιπρόεδρος Ταρκόφσκι την επόμενη Δευτέρα, 11 του μηνός, να συζητήσει τους ε, πολινούς βουλευτές της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων της Πολωνίας που θα επισκεφθούν για δύο μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι παρόν, ο Ταρκόφσκι θα με ε, αντικαταστήσει. Φυσικά όποιος όπως σας θέλει να είναι παρόν στη συνάντηση αυτή, αυτό θα είναι ικανοποίηση και για τους Πολωνούς συναδέλφους και για την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Πέρα των εργασιών.